Okay, Συγγνώμη, δεν έχουμε πάρα πολλά μέλη, είναι αλήθεια. Αλλά η συνεδρίαση αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο, οπότε μπορεί να την παρακολουθούν και να επανέλθουν αργότερα. Στα πλαίσια λοιπόν της νέας οδηγίας, για τις καταχρήσεις στις αγορές, τα θέματα MAD και MAR, έχουν γίνει κάποιες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οποίες θα σχολιάσουμε να αντιμετωπίσουν με σωστό τρόπο τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές και να προσπαθήσουμε να δούμε την ανεπάρκεια των ισχυουσών οδηγιών. Γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στη Μακάρτιν, η οποία είναι εισηγήτρια από πλευρά του Κοινοβουλίου για τα συγκεκριμένα θέματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε τόσους σημαντικούς εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά. Θα μοιραστούμε τις απόψεις τους και δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά. Νομίζω ότι θα ήθελα η σημερινή συνάντηση να είναι μια διαδικασία μαθητείας για μας σε σχέση με τις καταχρήσεις της αγοράς και τα insider dealings. Έχουμε μια οδηγία πάνω σε αυτό και αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να την αναθεωρήσουμε και να την μετατρέψουμε σε κανονισμό, κάτι το οποίο έχει λογική. Τα θέματα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε τα συζητήσαμε μάλλον σε μια συνάντηση και κλεισμένο των θυρών με τους εμπειρογνώμονες και σε κάποιες χώρες έχουν ήδη πάρει τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις έχουν ε, πράγματι θεωρήσει πολύ θετικές και ενσωματώσει. Ποινικέ κυρώσεις σαν παράδειγμα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει Μόνο τέσσερις χώρες στον τομέα αυτό έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν διώξεις και οι αστυνομικές αρχές ε, αναλαμβάνουν τις διαδικασίες αυτές, κάτι το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση αποτελεσματικό στις περισσότερες περιπτώσεις. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η οδηγία είναι λειτουργική. Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να σκληρύνουμε σε εισαγωγικά το σύνθημα είναι ότι το πλαίσιο παραβίασης των κανόνων της αγοράς είναι βασικό στοιχείο της μεταρρυθμιστικής ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να βρίσκουν τα κεφάλαια, να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογικούς τρόπους πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, Ξέρουμε ότι μέσω ακριβώς των τεχνολογικών βημάτων έχουν πολλαπλασιαστεί οι δυνατότητες για παραβιάσεις των κανόνων πρόσβασης σε χρήμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνο περισσότερες παραβιάσεις και καταχρήσεις, αλλά κυρίως πολύ πιο περίπλοκες μορφές καταχρήσεων και πολύ πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες μορφές καταχρήσεων. Αυτή είναι η άποψη λοιπόν της ομάδας μας, αυτή είναι η διαπίστωση που κάνουμε. Πρέπει να έχουμε ένα πεδίο ίσων ευκαιριών. Ξέρετε ότι πολλές φορές οι αγορές είναι σε ανταγωνισμό η μία με την άλλη και δεν θα πρέπει στη μία αγορά να υπάρχει μεγαλύτερη υπευθυνοποίηση σε σχέση με την δίωξη των παραβάσεων από ό,τι σε άλλες, γιατί αυτό στρεβλώνει γενικά τον ανταγωνισμό. Δεν θα περάσω λοιπόν στις λεπτομέρειες του περιεχομένου των μεμονωμένων αλλαγών οι οποίες προτείνονται. Ξέρω ότι τα μέλη θα ενημερωθούν μόνα τους σε σχέση με αυτό. Θα ήθελα όμως να σημειώσω κάποιες βασικές ε, αλλαγές, να υπογραμμίσω τις βασικές αλλαγές τις οποίες θέλω να επανέλθουμε. Um, measures to improve the prevention and detection of market abuse, measures to ensure public Λοιπόν, εδώ ε, προβλέπονται μέτρα και προτάσεις σχετικά με την καταγγελία των διαπιστώσεων αυτών, ακόμα και από πρόσωπα που δεν, έχουν άμεσο, δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενα, το θέμα των κυρώσεων, το θέμα της δημοσιοποίησης των παραβιάσεων. Έχουμε ήδη ε, δει ότι σε ορισμένες χώρες έχουν ενσωματωθεί τέτοιου είδους μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία. Καλωσορίζουμε επίσης ότι περιλαμβάνονται εδώ και οι ανταλλαγές ποσοτήτων, ανταλλαγές ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα. Είναι βασικό να συνεργαστούμε και με τον κύριο Φέρμπερ έτσι ώστε οι προτάσεις μας να είναι πλήρως συνακτικές και να αποφύγουμε θα έλεγα οποιαδήποτε περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού μέσω των ρυθμίσεων που ισχύουν σε κάθε χώρα και να αποφύγουμε επίσης και οποιαδήποτε μορφή αρμπιτράζ διαιτησίας ανάμεσα στις αγορές μέσω των ρυθμίσεων που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα ήθελα απλά να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να καταλάβουν καλύτερα τις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ λοιπόν Αρλίν. Καλωσορίζω τους ομιλητές μας το πιο απλό είναι να σας ζητήσω να πάρετε το λόγο στη σειρά που έχετε ε, καταγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Προσπαθήστε όμως παρακαλώ να σεβαστείτε ε, τα πέντε λεπτά τα οποία έχετε στη διάθεσή σας. Ακόμα και αν έχετε 7 λεπτά πρέπει να μειώσετε λίγο το κείμενό σας, την παρέμβασή σας. Δεν μπορείτε να μιλάτε πιο γρήγορα εξ αυτού γιατί η διερμηνία δεν θα σας ακολουθήσει. Προσπαθήστε λοιπόν παρακαλώ να σεβαστείτε τον χρόνο σας και να μην μιλάτε ταυτόχρονα πάρα πολύ γρήγορα. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Guy Sears, ο οποίος έγινε εκπρόσωπος του International Investment Management Association. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής που με καλέσατε εδώ. Η Investment Management Association αντιπροσωπεύει ε, διευθυντές ε, περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων και κεφαλαίων που ανήκουν σε διάφορα συνταξιδοτικά ταμεία, ε, σε επενδυτές λιανητής, σε κεφάλαια θα πρέπει να δρούμε προς το καλύτερο συμφέρον των πελατών μας και να έχουμε υψηλά πρότυπα εκτέλεσης μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και έντιμοι. Εμείς θέλουμε οι μεσίτες τους οποίους χρησιμοποιούμε τις αγορές όπου προσδιορίζονται οι τιμές, όπου ανακαλύπτουμε τιμές και οι εταιρείες τις οποίες επενδύουμε να έχουν επίσης υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς και εντιμότητας. Γι' αυτό τα μέλη μας έχουν δεσμευτεί να ακολουθούν ένα αυστηρό καθεστώς σχετικά με την κατάχρηση αγοράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, δεν, έχουμε, δεν κατέχουμε απλώς ε, ε, μετοχές ή χρέος των εταιριών. Πολλοί έχουν συνεχή διάλογο με την ανώτερη δίκηση των εταιριών για να θέσουν ερωτήσεις και και όπως ξέρετε, ε, το Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αναθεωρούν και ε, εξετάζουν ε, την διακυβέρνηση την εταιρική σε πάρα πολλά θέματα ούτω ώστε ε, για να και υπάρχει μια ε, πρόταση σχετικά με το γεγονός ότι βασιζόμαστε πάρα πολύ σε βαθμολογήσεις ε, και αξιολογήσεις. Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής υποστηρίζουμε την συμπερίληψη μέσων που είναι δεκτά στις συναλλαγές σε ρυθμισμένες αγορές. Επίσης, ε, έχουμε ρυθμισμένε αγορές και προϊόντα που είναι αντικείμενα συναλλαγής. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ψεύδο αγορά ε, με το να συναλλασσόμεθα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες που επεκτείνονται σε μεγάλο ε, έδαφος. Επίσης έχουμε την Αυστριαλιανή αγορά ε, και βλέπουμε αν υπάρχουν εκεί προϊόντα τα οποία είναι αντικείμενα συναλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουμε προτάσεις που είναι στη ΜΥΦΙΔ, στην οδηγία δεν ξέρουμε ποιο, θα είναι το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος OTF και τι θα θεωρούνται OTF και ποια θα είναι όλα τα μέσα τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών. Δεν ξέρουμε αν οι προτάσεις θα είναι ανάλογες με όλα αυτά τα δυνατά, τα εφικτά μέσα. Εκεί ενώ ε, η OETF είναι ένα προϊόν μετοχικό θα θέλαμε να καλύπτονται αυτά τα πρότυπα. Θα πρέπει διότι οι μετοχές οι οποίες αποτελούν αντικέμενο συναλλαγών ε, πρέπει να, ε, να ανταλλάσσονται σε μια ρυθμιζόμενη αγορά ή σε OETF. Θα θέλουμε να μην υπάρχει γραφειοκρατία για όλες τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει χειραγώγηση μετοχών επειδή οι μετοχές ανήκουν σε έναν εκδότη που είναι από μικρομεσαία επιχείρηση σχετικά με την εσωτερική πληροφόρηση και την διευρυμένο ορισμό. Νομίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτές αλλά που θα απαγορευθούν. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην μπούμε ανέφικτο, για τις εταιρείε διαχείρισης ε, διαθεσίμων να έχουν ε, επιχειρήσεις όπου υπάρχουν μεσίτες και ανώτερη δίκηση και διαχειριστές που έχουν τέτοια πληροφόρηση. Δεν ξέρουμε αν αυτά είναι σχετικά ή μη σχετικά σε σχέση με τους επενδυτές. Επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο πώς κανείς μπορεί να ξεπληθεί από αυτήν την πληροφόρηση αν τη χρησιμοποιήσει εφόσον η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να την δημοσιοποιήσει. Έχουμε πάντοτε υποστηρίξει την προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν λέμε ότι πρέπει να είναι η προσέγγιση της Ευρώπης, αλλά υπάρχει μια ισοδύναμη πρόταση και μια και η δική μας πρόταση το αναφέρει αυτό. Το υποστηρίζουμε αυτήν την συμπεριφορά, αλλά στην χρήση στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένας χαρακτηρισμός ότι ε, δηλαδή η συμπεριφορά της διάδοσης της πληροφορίας μπορεί να θεωρηθεί ως αποτυχία από το ενδιαφερόμενο άτομο να τηρήσει τα πρότυπα και τους κανόνες συμπεριφοράς ε, που αναμένονται θα μπορούμε να χάσουμε το άρθρο 6.1 ε που είναι σχετικά με την σχετική εσωτερική πληροφόρηση. Διότι όσα είναι σχετικά ε, δεν μπορούν όλα να χρησιμοποιηθούν και για να δούμε τι πρέπει να κάνει μια χώρα η περίπτωση Spector, γνώση και αιτίες. Δεν ξέρουμε αν η χρήση πληροφόρηση είναι συναλλαγή βάση της πληροφόρησης ή συναλλαγή όταν κανείς κατέχει την πληροφορία. Θα πρέπει να δούμε ένα άτομο αν δρά βάση της πληροφόρησης, όχι μόνο αν κατέχει την πληροφόρηση, αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφείς, διότι αυτό δεν παρεμποδίζει μια συναπόφαση ότι δηλαδή ένα άτομο που είχε την πληροφόρηση αν όντως την χρησιμοποίησε. Νομίζω τα τεκμήρια θα πρέπει να αναφέρονται. Ε, νομίζουμε ότι ε, το κινέζικο τείχος είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις για να μειωθούν οι κίνδυνοι διαρροής πληροφοριών και οι επόπτες θα πρέπει να εξετάσουν τα συστήματα και τους ελέγχους HFT. Βεβαίως θα το θεωρήσουμε αυτό. Δεν, Δεν ξέρουμε αν υπάρχει ανάγκη να το προσδιορίσουμε αυτό και αν πρέπει να το συζητήσουμε. Υπάρχουν μερικά ασφαλή καταφύγια στην οδηγία τα οποία δεν επαναλήφθηκαν στην πρόταση βάσει ανάλυσης δημοσίων στοιχείων και νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Ξέρω ότι πέντε λεπτά δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και ίσως μήπως θα, όταν θα έχουμε την συζήτηση και τις ερωτήσεις θα θέλετε να προσθέσετε κάτι. Έχουμε τώρα από την επενδυτική τράπεζα BNP Paribas, τον κύριο Βαλόνσα. Είναι μια επενδυτική τράπεζα για τις προτάσεις ΜΑΡ και ΜΑΤ, διότι υπάρχει ανάγκη να συμπληρώσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνοντας το μεγάλο φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων όπως είναι τα εμπορεύματα ε, και επίσης να λάβουμε υπόψη το MTF και τα OTFs. Ένα θέμα θα είναι ο καλύτερος συντονισμός, εποπτεία του spot market που συνήθως ρυθμίζονται από διάφορες οργανώσεις ανάλογα με τη χώρα και την δικαιοδοσία σχετικά με τις κυρώσεις και την εφαρμογή. Υποστηρίζουμε την εφαρμογή, την επιβολή ε, μέτρων ε, δεσμευτικών. Αυτό και τις κυρώσεις ε, της ε, διοικητικές. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να έχουν άμεση εξουσία πραγματική να λαμβάνουν μέτρα διοικητικά και επιθαρχικά, χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται σε δικαστήρια είμαστε πιο προσεκτικοί όσον αφορά ε, στην αναθεώρηση των catch-all concepts. Σχετικά με την εσωτερική πληροφόρηση, ξέρουμε ότι η πρόταση σχετίζεται με παράγωγα, ε, με εμπορεύματα και με διάφορες ε, εκδόσεις αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη την αντίληψη της πληροφόρησης που είναι σχετική αλλά δεν είναι δημόσια διαθέσιμη. Πρέπει να διευρύνουμε την έννοια της εσωτερικής πληροφόρησης πράγμα που θα έχει επιπτώσει στα εσωτερικά συστήματα παρακολούθησης και εποπτείας και στις διαδικασίες των επενδυτικών εταιριών. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει αυτού του είδους η πληροφόρηση που είναι ευαίσθητη να ληφθεί υπόψη. Έχουμε επίσης ένα θέμα με ευρύτερη, ευρύτερο ορισμό της φυραγώγησης αγοράς που συμπεριλαμβάνει την έννοια της συμπεριφοράς. Θα θέλαμε η έννοια της συμπεριφοράς να προσδιοριστεί καλύτερα στην οδηγία. Δεν έχουμε κανένα θέμα σχετικά με την έννοια του attempt ε, του εγχειρήματο της προσπάθειας, ε, διότι εκεί αναφερόμεσα ε, στον ρυθμιστή σχετικά με τα ασφαλή καταφύγια, τα οποία ήταν στην πρώτη οδηγία το, η ρευστότητα του παρόχου που υπάρχει σε ορισμένα δίκαια στην Γαλλία και που μια, θεωρείται σαν μια αποδεκτή πρακτική της αγοράς για την εξασφάλιση ρευστότητα για μετοχές, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα θέλαμε ε, τις, ε, τους κανόνες pre-marketing που σήμερα δεν έχουν εναρμονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποτελέσουν μέρος της οδηγίας κατάχρησης αγοράς διότι έτσι ε, θα είναι ίση η όρη και αυτό είναι καλό για την την πρωτογενή αγορά. Θα ήθελα να κλείσω σχετικά με το, τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Ε, δεν είναι, ονομαζόταν αρμπιτράζ πριν από 20 χρόνια, αλλά η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας με ε, ε, με ορισμένα στόπους που είναι ε, συνέπειες της οδηγίας MIFID 1 έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αλγοριθμικού αρμπιτράζ και υπάρχουν πάρα πολλές στρατηγικές επιθετικές όπως είναι το single stock arbitrage, όπως το arbitrage που βασίζεται σε δείκτες ή σε πανέρια δικτών Υπάρχουν επίσης διάφοροι ε, πρωταγωνιστές. Έχουμε ρυθμιζόμενες ε, τράπεζες, ε, επενδυτικές εταιρείες σε σχέση με κεφάλαια που δεν είναι καταχωρημένα με διαφορετικά επίπεδα διαφάνειας στις δραστηριότητες τους. Βεβαίως, για τις, έχουμε διαφάνεια για τις τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την ρευστότητα στην αγορά για την καλή λειτουργία και την μείωση των απειλών και κινδύνων. Αν έχουμε επαγγελματίες που υπόκεινται σε ρυθμίσεις και καλή παρακολούθηση και εποπτεία, Έχουμε, μπορούμε να αναφερθούμε στην ΣΥΦΜΑ που είναι μια οργάνωση της, των Ηνωμένων Πολιτειών και την μελέτη AMF. Δεν υποστηρίζουμε την ιδέα των τεχνητών περιορισμών ή της απαγόρευσης. Υποστηρίζουμε την ιδέα να υπάρχει μια ειδική άδεια για τις εταιρείε που έχουν ε, συναλλαγές με μεγάλη συχνότητα ε, ακόμα και κεφάλαια, κεφάλαια που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Ο ρυθμιστής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείε είναι καλά εξοπλισμένες ε, για την εποπτεία, την παρακολούθηση, για να αποφευθεί κάτε, κατα, κατάχρηση ή δυσμενής επίπτωση στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια περνάμε στα θέματα 1 και 2 και νομίζω έχει αυτό προσαφινιστεί. έχουμε τον επόμενο Γενικό Διευθυντή, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και εισηγητή για την κατάχρηση θέσεως αγοράς και που θα λάβει τον λόγο αμέσως στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητή, αγαπητή εισηγητά. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι παρόν, να, παρουσιάσω κάποιες σκέψεις όσον αφορά την κατάχρηση αγοράς. Οι κανόνε για την αντιμετώπιση κατάχρηση θέση στην αγορά είναι θεμελιώδου σημασία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Είναι όμω ε, μια ε, αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη. Αφενό πρέπει να έχουν καλώ σχεδιαστεί αυτέ οι προτάσει ε, αναλογικά ώστε να αποφεύγονται ερμηνευτικές ή άλλες εφαρμοστικές διατάξεις και να είναι και αποτελεσματικές. Από την άλλη πλευρά πρέπει να συμπληρώνονται να συμπληρώνονται με αποτελεσματική εποπτεία. Σε σχέση με την οδηγία για να την η κατάχρηση θέση στην αγορά, θα πρέπει σε σχέση με τι εσωτερικέ πληροφορίε αμέσω να δρούμε. Δηλαδή, του ίδιου τύπου πληροφορίε, insider information, να είναι η βάση για την απαγόρευση καθώ και για την υποχρέωση αποκάλυψη. Αυτή η σύμπτωση ενιών δημιούργησε πάρα πολλέ νομικέ αβεβαιότητε, ιδιαίτερα επειδή η κατάχρηση θέση στην αγορά ήταν ήδη η βάση για την έναρξη διαβημάτων και δράσεων για την δίωξη σε κράτη-μέλη. Υπήρξε περιορισμό ε, για το ότι δεν θα έπρεπε τέτοιου είδου ε, διορίε να είναι παραπλανητικέ. Για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, πολλά κράτη-μέλη δεν εφάρμοζαν απλά την οδηγία ή την παράκαμπταν με κατευθυντήριε γραμμέ ε, των ίδιων, των ίδιων υπεύθυνων αρχών όμως ήταν πραγματικά άχρηστες όταν είχαμε θέματα εγκληματικών ε, κατηγοριών. Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια το σχέδιο κανονισμού έχει το προτέρημα να αναγνωρίζει ότι χρειάζεται μια διαφοροποίηση. Και έτσι διαφοροποιούμε, διαφοροποιούμεθα σε σχέση με, την πληροφορία, με τις πληροφορίες ε, που δεν μπορεί να τύχουν ε, κατάχρησης. Αλλά γίνεται αυτό με λάθος τρόπο. Σε σχέση με την μη κατάχρηση εσωτερικών πληροφοριών εισάγεται ένα νέο άρθρο το 6ε που είναι σχετικό μόνο σε περιπτώσει κατάχρηση. Δεν τεθεί ποτέ σε διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εισάγει μια νέα φάση για τι ε, εσωτερικέ πληροφορίε ε, που επικεντρώνονται σε ένα αυστηρό φάσμα αυτών των θεμάτων όπω είναι γνωστό μέχρι σήμερα αλλά το παράδειγμα το υπόδειγμα είναι διαφορετικό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι δεν υπάρχει επάρκεια όσον αφορά την, ε, τους σαφείς ορισμούς. Θα πρέπει να περιγράφεται σαφώς η παραβίαση και να μην αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των δικαστηριών για να επιτρέπεται οι πολίτες να κατανοούν εύκολα αν έχει κάνει κάποιος μια τέτοια παράβαση ή όχι και η διεύρυνση του καταλόγου σε σχέση με τις δυνατότητες ε, δίωξης ε, θα πρέπει να μην μας οδηγήσει στην, ε, περιορισμό της ρευστότητα. Επίσης, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τους μεριδιούχους. Αν υπάρχει περιορισμός για τις αρμοδιότητες τους σε σχέση με τις συναλλαγές τους. Δύο, λοιπόν, κύριες αλλαγές είναι αναγκαίες. Το νέο αυτό άρθρο πρέπει να διαγραφεί. Πρώτον. Δεύτερον, η αποκάλυψη των πληροφοριών στο άρθρο 12 πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον παλαιό ορισμό για τις ε, πληροφορίες εκ των ένδων. Εν πάση περιπτώσει η απέτηση για έναν κατάλογο που πρέπει να μην οδηγεί σε παραπλάνηση των πολιτών σε σχέση με την χρήση ε, των ένδων πληροφοριών, πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο να εφαρμόζεται, πρέπει να δίνει την δυνατότητα να αποκαλύπτονται στοιχεία σε σχέση με διαβουλεύσεις από τις επιχειρήσεις μόνο όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος βαθμός βεβαιότητας έτσι βλέπουμε ότι χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 29 και το 30 της οδηγίας όπως προαναφέρθηκε δηλαδή ο συνδυασμός αυτών των δύο αποκλείει τις πληροφορίες ε, όσον αφορά και την πρόθεση εσκεμένα να αποκαλύπτονται στοιχεία και τα δύο αυτά στοιχεία πρέπει να επανεισαχθούν στον κανονισμό πιθανόν στο άρθρο 6 για τις φήμες είναι ένας, ε, ε, μια σαφής περίπτωση που ούτε στο σημερινό σχέδιο πρότασης ε, εμπεριέχεται. Όταν δηλαδή έχουμε το πρόβλημα να συμπεριφερθούμε σωστά όταν αντιμετωπίζουμε φήμες και ψιθύρους. Δημιουργείται αβεβαιότητα, ανασφάλεια, διότι αυτή η διασπορά φήμων μπορεί να οδηγήσει σε μια πλήρη παραπλάνηση εταιριών το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να στέλνει ή να προσπαθεί να στείλει τέτοιου είδους ε, μηνύματα μπορεί να εξισούται με παραβίαση σε σχέση με τον εκδότη καλύτερο θα ήταν να μην αποκαλύπτονται τέτοιες πληροφορίες αντί να υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης παραπλανητικών πληροφοριών. Θα, μπορούσε να θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε λιγότερη πληροφόρηση για τους επενδυτές. Θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό μόνο τότε να σχολιάζουν οι εταιρείε όταν υλοποιούνται δύο προϋποθέσεις. Όταν είναι αληθής η φήμη και όταν υπάρχουν ανώμαλες κινήσεις σε σχέση με τον όγκο των συναλλαγών. Διαφορετικά δεν θα έπρεπε καμία τέτοια προσέγγιση να ακολουθείτε. Όσον αφορά την ε, διαβούλευση θα πρέπει να απαιτείται όταν έχουμε ένα κατόφλι το οποίο υλοποιείται. Ο υπολογισμό του κατοφλίου θα πρέπει να ξεκινά από το μηδενικό επίπεδο μέχρι ότου φτάσουμε την τιμή αυτού του ε, κατοφλίου. Μία τέτοια πληροφόρηση, ειδοποίηση πρέπει να αποστέλλεται από τους ε, αρμόδιους μιας εταιρείας στις αρμόδιες αποκλειστικά αρχές. Ένα, μια περίπτωση που μπορεί να αποστελλεται απο τους αρμοδιους μιας εταιρειας στις αρμοδιες αποκλειστικα αρχες μια περιπτωση που μπορει να εξισωθεί με το short selling. Και μπορούμε να πούμε ότι ε, από πέντε ημέρε, σε δύο ημέρε ε, συντέμνεται, πράγμα το οποίο μπορεί να συνεπάγεται δυσκολίε Σε σχέση με την χρησιμότητα, τουλάχιστον όσον αφορά τι ε, εταιρείε. θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλε τι εταιρείε αυτή η ενημέρωση, τουλάχιστον σε όλε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, οπουδήποτε και αν γίνεται η συναλλαγή. Τελευταίο σημείο, η υποχρέωση τη αποκάλυψης των πληροφοριών και των στοιχείων αυτών όσον αφορά εναλλακτικέ αγορέ και δράσει. Αυτό δεν είναι εύθετο. Η απλούστευση όσον αφορά την ε, αντιμετώπιση κατάχρηση θέση στην αγορά, εταιρείε καθώς επίση ε, και η απαρίθμηση των περιπτώσεων αυτών ενδιάμεσα δεν θα πρέπει να ε, καλύπτονται οι πιθανοί επενδυτές. Αυτοί θα πρέπει με συνεπή τρόπο να φέρονται με και την επιβολή των κανόνων αποκάλυψης θα περιορίζαμε τις δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διεκδίκησης των κεφαλαίων τους. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί αυτή η μορφή αυτών των ρητρών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να σας ε, υπενθυμίσω όταν διαβάζετε ακολουθείτε πολύ ταχύτερο ρυθμό από ότι όταν ομιλείτε φυσιολογικά. Κάνουν εξαιρετική δουλειά οι διερμηνείς αλλά να μην μιλάτε με τέτοιο ταχύτατο ρυθμό. Patrick στη συνέχεια σύμβουλος των οικονομικών αγορών και ε, εμπειρογνώμων στα θέματα χρηματοδότησης FME. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερη χαρά να είμαι παρόν εδώ σήμερα, να προσφωνήσω τα μέλη της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής και να συζητήσω το πολύ ενδιαφέρον θέμα όχι μόνο της κατάχρησης θέσης στην αγορά, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πραγματικά φτάσαμε πλέον ένα θαυμάσιο νέο κόσμο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10-15 ετών όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο και αυτό άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το πώς λειτουργούν όλες οι χρηματοοικονομικές αγορές. Ταυτόχρονα έγινε πολύ ενδιαφέρον αυτό ως διαδικασία διότι ανοίγει η ευκαιρία για έναν Τελείω καινούριο κόσμο όσον αφορά την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις συναλλαγέ. Και προ αυτόν τον στόχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τύχουν συγχαρητηρίων για την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα λειτουργίας. Οι παρατηρήσει μου αφορούν τι τις επιχειρήσει. και όχι μόνο αυτές τις αγορές ε, που έχουμε ήδη σήμερα όπως ε, το χρηματιστήριο της Βασοβίας όσον αφορά την κεντροανατολική Ευρώπη αλλά και σε σχέση και με την ε, καταχώρηση ε, επιτυχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στρεφόμεθα όμως και στις ε, μικροκεφαλαιακές συναλλαγές από πλευράς επιχειρήσεων και των πολύ μικρών αγορών που μπορούν να καλυφθούν με το διαδίκτυο σήμερα. Ξέρουμε ότι το νομοθέτημα Μακένρι στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε την δυνατότητα να ξεκινούν με ένα εκατομμύριο τέτοιες επιχειρήσεις και με ταχύτατο αριθμό να υποστηρίζονται και εταιρείε ε, με κεφάλαιο κίνησης 2 εκατομμυρίων. Πρέπει να δούμε ε, εκ του σύνεγγυ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές χρειάζονται ένα πιο ελαφρύ, εύκαμπτο ρυθμιστικό πλαίσιο. Θέλω να τονίσω ότι αυτό βέβαια δεν σημαίνει απουσία ρυθμιστικού πλαισίου. Σημαίνει λειτουργία σε ένα θεσμικό πλαίσιο ρυθμιστικό που θα είναι λειτουργικό και δεν θα προσθέτει υπερβολικό βάρος αριθμίσεων και διατάξεων στις επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν σε τέτοιε συναλλαγέ. Όσον αφορά αυτό, πιστεύω ότι όπω και σε άλλε τέτοιε καταχωρήσει, η ιδέα για το σημερινό MTF ε, είναι μια πολύ υγιή ιδέα και αξιόπιστη. Θέλω όμως να επικεντρωθούμε και σε ένα συγκεκριμένο ενιαίο σημείο ρύθμισης και με συγκεκριμένα στοιχεία για την καταχώρηση ώστε πάντα να μπορεί να αξιολογείται αμέσως η περίπτωση κατάχρησης θέσεως στην αγορά αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πράγματι η απλούστευση του νέου πλαισίου μικροσυναλλαγών, micro exchange, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, είναι ότι η ιδέα πρέπει να είναι να έχουμε ένα μητρό με μικρότερες, λιγότερες ε, περιτές ε, διατάξεις και επιβαρύνσεις όσον αφορά για τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται Και γενικότερα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ένας μεγάλος βαθμός των λειτουργιών αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι η καταχώρηση και η καταχώρηση των στοιχείων του αυτών αντί να παράγεται μια ολόκληρη γενεά στοιχείων όπως συμβαίνει με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και εταιρείε που καταχωρούνται στα χρηματιστήρια. Φτάνουμε σε ένα σημείο που εξετάζοντας την σταδιοδρομία μιας μικρής μικρομεσαίας επιχείρησης πρέπει να δούμε ένα χαμηλού επίπεδου ρυθμιστικό πλαίσιο απαιτήσεων όσον αφορά τις επιβαρύσεις και Καλωσορίζουμε την ιδέα αναλογικά να υπάρχει επιβάρυνση ανάλογα με τον όγκο αυτών των επιχειρήσεων. Διότι σίγουρα χρειάζονται χρηματοδότηση αυτέ οι επιχειρήσει, χρειάζονται εναλλακτικέ πηγέ χρηματοδότηση, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζε αντιμετωπίζουν προβλήματα μόχλευση. Ιδιαίτερα εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω πολίτε χρειαζόμαστε να έχουμε το δυνατόν περισσότερε ευκαιρίε να ιδρύονται τέτοιε επιχειρήσει στο μέτρο του εφικτού. Η ε, ιδέα λοιπόν μια ενιαία ε, ρύθμιση για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ζωτική σημασίας, καθώς θα είναι μια σχετική, πιο, ε, μια σχετική διευκόλυνση, ελαφρύτερη επιβάρυνση και όταν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γίνουν μετά από ρήμανση μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα μπορούν να προχωρήσουν σε άλλου είδους καταχωρήσεις όπως στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ή την Nasdaq ή άλλων τέτοιων θεσμικών οργάνων εξ ονόματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αυτό πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική προοπτική. Σας ξαναδίνω λοιπόν το λόγο, ολοκλήρωσα κάτω από πέντε λεπτά πρόεδρε, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσω τώρα στην κυρία Φων Χάρτμαν υπεύθυνη της uh, Nasdaq περιοχή Βόρειας Ευρώπης. Γεια σας, ε, λέει η κυρία Φων Χάρτμαν. Είναι τιμή μου για μένα που είμαι εδώ σήμερα. Το Nasdaq, ο MX ασχολείται με τις αγορές ομολόγων στις Βαλτικές, τις Βόρειες, Σκανδιναβικές χώρες και την Ισλανδία. Στις 7 ε, αγορές κάνουμε λίστες και συμπεριλαμβάνουμε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και προϋπόθεση για να λειτουργήσουν οι αγορές είναι φυσικά η εμπιστοσύνη. Εκτός από την Ισλανδία η επίβλεψη των αγορών γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο, είναι συγκεντρωμένη θα έλεγα η μορφή ελέγχου στο κέντρο. Οι σκανδιναβικές χώρες είναι η δική μου ευθύνη, η πραγματική επίβλεψη συγκεντρώνεται στη Σουηδία, αν κάτι ανοιχνεύεται το σχετικά ύποπτο, φυσικά γίνονται έρευνες και σε τοπικό επίπεδο ε, γίνονται ε, θα έλεγα διαδικασίες και σε σχέση με την νομοθεσία σχετικά με τις ύποπτες συναλλαγές και οι αναφορές ε, μεταφέρονται επίσης και ανακοινώνονται και στην τοπική ρυθμιστική αρχή. Αυτό περιλαμβάνει και προϊόντα και γενικά αγορές της Νορβηγίας αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου μερικές φορές. Πιστεύουμε ότι η επίβλεψη, η εποπτεία καλύτερα είναι βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της αγοράς. Δεν θεωρούμε ότι είναι ένα κόστος το οποίο θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε. Αντίθετα, η εποπτεία είναι ένα πλεονέκτημα. Είναι κάτι το οποίο προσδίδει αξία στην τοπική αγορά. Είναι κάτι το οποίο συνεισφέρει στην δίκαιη και ε, θα έλεγα διατεταγμένη λειτουργία της αγοράς και φέρνει εμπιστοσύνη στις αγορές. αλλά θέλουμε να είμαστε φυσικά πιο αποτελεσματικοί. Η εποπτεία σε πολλές αγορές ταυτόχρονα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια των ολοκληρωμένων αλλά και πολυδιασπασμένων πολλές φορές αγορών. Έχουμε κάνει αρκετά, θέλουμε όμως και περισσότερα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την εναρμόνιση της επιβολής και των κυρώσεων είναι κάτι το θετικό δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές στην Ευρώπη λόγω τοπικών ασθενέστερων ρυθμίσεων. Αλλά επειδή τα δικαστικά συστήματα στην Ευρώπη είναι διαφορετικά, δεν μπορούμε να φτάσουμε δυστυχώς ή ευτυχώς στο 100% εναρμόνιση. Το βασικό μας πρόβλημα όμως είναι η ανείχνευση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της σα θα έλεγα, ρύθμισης είναι ακριβώς η αδυναμία ανείχνευσης μερικές φορές σε μια πολύ διασπασμένη αγορά και εδώ αναφέρομαι και στην ε, MAD, την Οδηγία για την Κατάχρηση στις Αγορές και τα MIFID. Πρώτον, σήμερα μια αγορά μπορεί να παρακολουθήσει την αγορά μέσα στην οποία λειτουργεί. Οι traders όμως δραστηριοποιούνται σε ε, μη πραγματικό χρόνο σε πάρα πολλές αγορές. Το σύστημα το οποίο λειτουργεί για συνεργασία ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές περιλαμβάνει φυσικά και ανταλλαγές εκθέσεων και καταλόγων συναλλαγών αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει κάποια μορφή real-time ε, ε, εποπτείας των εντολών αγορών, δεν καλύπτει όλα τα κενά. Και γι' αυτό μπορούν να υπάρξουν κάποιες καταχρήσεις ε, χωρίς να ανοιχνεύονται σε πραγματικό χρόνο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το MIFID 2 αναγνωρίζει το πρόβλημα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Έχοντας συζητήσει το θέμα αυτό και με τα χρηματιστήρια και με τις ε, επιχειρήσεις και με τα MTFs, ε, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Η πρωτογενής αγορά για κάθε ε, κομμάτι, σαν παράδειγμα το Ελσίνκι για την Όκια, σαν παράδειγμα, θα πρέπει να ορίζεται υπεύθυνο για κάθε συναλλαγή στον συγκεκριμένο χώρο της αγοράς αυτής. Η πρωτογενής αγορά είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπενευθυνοποιούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, γιατί είναι σε μόνιμη σχέση και διάλογο με όλους τους εκδότες μετοχών. Νομίζω ότι ο έλεγχος όλων των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο θα βελτιώσει την ανείχνευση των καταχρήσεων. Η τεχνολογία δεν είναι πρόβλημα. Υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να παρακολουθούν πολλές αγορές ταυτόχρονα από τον ίδιο χώρο. Όπως είπα, εμείς στο Nasdaq OMX έχουμε ήδη συγκεντρώσει την εποπτεία μας σε επίπεδο πραγματικού χρόνου. Για να το πετύχουμε πλήρως αυτό, καταρχάς ορίζουμε την πρωτογενή αγορά σε κάθε περίπτωση, ζητάμε από όλες τις αγορές να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να απομακρυνθούν πρέπει όλα τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών κατανέμουμε εκ των προτέρων το κόστος της διαδικασίας εποπτείας και θα πρέπει να ανταλλάσσονται φυσικά ανάμεσα στις αγορές οι απαραίτητες πληροφορίες. Φυσικά θα πρέπει να περιορίζεται η χρήση των δεδομένων τα οποία μεταφέρονται για λόγους εποπτείας και όχι για άλλους εμπορικούς λόγους. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτά για άλλου είδους εμπορικές πραγματικά δραστηριότητες όπως ε, δεν ε, είχε ξεκαθαριστεί σε επίπεδο ΜΥΦΙΔ 1. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι νομοθέτες ε, ήταν πολύ αυστηροί σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο καλούμεθα να οργανωθούμε. Πάντως απαιτείται να βελτιωθεί η ανταλλαγή των δεδομένων και ποσοτικά και ποιοτικά. Η ποσότητα είναι ικανοποιητική, αλλά η ποιότητα πρέπει να βελτιωθεί. Οι αρχές εποπτείας πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν συγκρίσιμα, αν θέλετε, στοιχεία. Αυτό θα βοηθήσει την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στις αγορές, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό μας πρόβλημα σήμερα. Η κατάχρηση της αγοράς είναι όλο και πιο επαγγελματική και οργανωμένη. Για να καταπολεμηθεί αυτή η κατάχρηση καλούμεθα να είμαστε επαγγελματίες και οργανωμένοι και σε επίπεδο σχεδιασμού και ρύθμισης και σε επίπεδο εποπτείας και σε επίπεδο επιβολής. Η επιβολή είναι κομβικό. Ε, αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την επιβολή πρέπει να έχουν τα μέσα να εφαρμόζουν άμεσα και αποτελεσματικά πέραν των τοπικών συνόρων τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα. Η πρόταση για μια οδηγία λοιπόν και για ποινικέ κυρώσεις φέρνει στην επιφάνεια το θέμα της ευθύνης των νομικών προσώπων, όπου κάποιος ο οποίος είναι ηγετικό τέλεχος σε μια επιχείρηση κατηγορείται για την ενέργειά του η οποία ήταν όμως προς όφελος του νομικού προσώπου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον νομικά και είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει στο μέλλον στη καταπολέμηση των καταχρήσεων των αγορών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τέλος έχουμε τον Ροτρίγκο Μπουεναβεντούρα ο οποίος προέρχεται από την ΕΣΜΑ, από την αρχή την Ευρωπαϊκή για τις ε, αγορές και τις εκδοσίες. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, για την αναθεώρηση σε σχέση με την πρόταση οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια και παγιώνει τα στοιχεία σε σχέση με την καλή του λειτουργία και προοδεύει σε άλλους τομείς όπου χρειαζόταν πρόοδος. Ένα στοιχείο κλειδί είναι η συμπερίληψη των περισσότερων κανόνων και κανονισμών στην ρύθμιση σε σχέση με έναν εναρμονισμό της αντιμετώπισης κατάχρησης θέσης αγοράς. Επικεντρωνόμενοι σε σχέση με την επιβολή και των κυρώσεων θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια συμπληρώνοντας τα άλλα θέματα. Στου ε, ορισμούς. Είναι θεμελιώδε να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες για την εποπτεία θα εφαρμόζονται σε, όλες, ε, σε όλα τα είδη των περιπτώσεων και θα ευθυγραμμίζονται με τους ορισμούς ε, MIFID. MIFID και MAD θεωρώ ότι συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους και είναι θεμελιώδους σημασία να συνεχιστεί αυτό. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις ε, αναφορές και εκθέσεις ε, για τις συναλλαγές ε, μέσα στο πλαίσιο MIFID πρέπει να χρησιμοποιούνται και για την εποπτεία αγοράς υποχρεωτικά. Δείχνεται ότι σε σχέση με την εποπτεία των πελατών με ενδιάμεση έκθεση αυτό είναι ένα στοιχείο παρακαλώ να επιβραδύνετε λίγο για να μην ταλαιπωρούνται οι διερμηνείς. Είναι ένα στοιχείο που σύμφωνα με τις χώρες εκείνες όπου συλλέγονται αυτά τα στοιχεία βελτιώνει σημαντικά την ε, ακρίβεια και την ποιότητα της εποπτείας ε, κατάχρησης της αγοράς. Τώρα είναι πιο κατακαιρματισμένες οι συναλλαγές ε, και πιο πολυσχηδείς από ότι το 2003 όταν εγκρίθηκε αυτή η προσέγγιση και αυτό απαιτεί θεμελιωδώς αλλαγές ε, στις, ε, στη μεθοδολογία για να ανοιχνεύονται τέτοιες περιπτώσεις κατάχρησης. Ωστόσο, δεν θεωρούμε ότι μια ριζοσπαστική ε, επαναδιάταξη χρειάζεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τα τρία επίπεδα ε, επιχειρήσεων, trading venues και επόπτες, εποπτικές αρχές μπορούν να συνεχίσουν να δρούν μέσα σε ένα σημαντικό πλαίσιο υπό τον όρο ότι θα ενημερώνονται και θα επικαιροποιούνται τα συστήματα και οι διεργασίες για να ανοιχνεύονται οι περιπτώσεις παραβιάσεων. Σε σχέση τώρα με το high trading, οι διατάξεις που ε, προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζονται για να προσαρμοστεί ο κατάλογος πρακτικών στο πλαίσιο συναλλαγών. Είναι εξίσου σημαντικό ο κανονισμός να μπορεί να επικαιροποιείται στο μέλλον μέσω ε, της διαδικασίας εντεταλμένων πράξεων ή της επικαιροποίηση ε, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θεωρούμε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές ΕΣΜΑ μπορούν να διαδραματίσουν και ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα στρέφομαι στις ε, αρμοδιότητες και εξουσίες των αρμόδιων αρχών. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε, πιστεύουμε, ότι η καταπολέμηση της κατάχρησης αγοράς απαιτεί ένα πλήρες σύνθετο πλαίσιο και γι' αυτό Καλωσορίζουμε την συμπερίληψη ρητά την πρόσβαση σε τηλεφωνικά και άλλα ηλεκτρονικά μητρώα και αρχεία, γιατί και αυτό είναι μια σημαντική πηγή για τις διακριβώσεις, ε, που στο σημερινό πλαίσιο όσον αφορά τις ε, τακτικές ε, και πρακτικές μας δημιουργεί κάποιες τριβές όσον αφορά και το καθεστώς προσωπικών δεδομένων. Είναι θεμελιώδου σημασία να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση σε τέτοιου είδους δεδομένα θα είναι δυνατό να εφαρμόζεται στην πρακτική εφαρμογή. Στις κυρώσεις καλωσορίζουμε την εισαγωγή κοινών κριτηρίων για τον καθορισμό κυρώσεων ιδιαίτερα για τον κοινό κατάλογο των επιλήψιμων πράξεων. Το ίδιο μπορεί να αναφέρουμε και για τις ελάχιστες ή και μέγιστες οικονομικές ε, πίνες και ε, πρόστιμα για να ε, για την αποφυγή οποιασδήποτε περίπτωσης arbitrage παρότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες πάντα και σε σχέση με την χρήση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων υπό το σημερινό πλαίσιο αναμένουμε ότι σύντομα θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και με ικανοποίηση θα μπορούν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από πλευράς μας. Σε σχέση με την εισαγωγή εγκληματικών τώρα ποινών για τέτοιου είδους παραβιάσεις και παραβάσεις κατανοούμε την λογική ότι πρέπει να αποσταλεί ένα σαφέστατο κάθετο μήνυμα στους πιθανούς ε, καταχραστές ε, τέτοιων πληροφοριών και τέτοια θέσης στην αγορά, ώστε να υπάρχει μήνυμα αποτροπής. Όταν όμως σχεδιάζουμε τέτοιου είδους διατάξεις πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι το ότι η γενικές ε, διοικητικές κυρώσεις από πλευράς των κρατών μελών, από πλευράς διοικητικού δικαίου είναι πολύμορφες και διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Και δεύτερον, Επόπτε για θέματα ασφάλεια σε πολλέ χώρε, σε πολλέ περιπτώσει έχουν αναπτύξει σημαντικέ δυνατότητε και ικανότητε από πλευρά συστημάτων και τώρα τα εφαρμόσουν όλα αυτά μέσω διοικητικών διαδικασιών για τις, ε, την δίωξη. Είναι λοιπόν σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι ο ορισμό ε, εγκληματικών περιπτώσεων ε, συμπεριφορά θα είναι συμβατό με την διατήρηση ενό διοικητικού πλαισίου και θα υπάρχει επαρκέ περιθώριο για του ρυθμιστέ να αποφασίζουν ποια οδό θα ακολουθήσουν την διοικητική, δικονομική ή την, ε, κατά, την δίωξη εγκληματική πράξεως ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει η πιο αποτελεσματική δράση σε σχέση με την εγκληματική δίωξη έναντι σε ε, αντιδιαστολή με την διοικητική δίωξη, αστική δίωξη για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ε, Είδα ότι οι να έχετε ερωτήσεις. Βεβαίως ε, προχωρούσατε πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως θα υπάρξουν ερωτήσεις. Ίσως και όδης. Ναι, θα ήθελα να θέσω ένα βασικό ερώτημα που αναφέρθηκε σε θέμα σε πάρα πολλές παρεμβάσεις και ίσως είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε ε, στην νομοθεσία. Ε, το θέμα αυτό της σχετικής ε, πληροφόρησης έχουμε το άρθρο 6.1 ε μήπως δεν θα συμφωνούσατε λόγω του επίπεδου πολυπλοκότητας και του επίπεδου ταχύτητας που έχουμε στο trading δεν ε, ίσως ε, θα μπορούσε να μας πει η BNP αν θα έπρεπε να έχουμε απαγόρευση, αν θα έπρεπε να δούμε ορισμένες πρακτικές που μπορεί να είναι καταχραστικές, ε, να δούμε ποιες είναι αυτές οι πρακτικές και χρησιμοποιώ το θέμα αυτό σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Ροντρίγκης από την ΕΣΜΑ. Πρέπει να έχουμε κάποια ευελιξία για τον ρυθμιστή, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πρακτικές οι οποίες είναι πολύπλοκες που καταχρώνται την αγορά και ορισμένες πρακτικές που όντως είναι καταχρηστικές. Ίσως θα πρέπει να έχουμε μια μελλοντική νομοθεσία αν προσπαθούμε να προσδιορίσουμε, να ορίσουμε κάτι αν είναι σχετικό ή δεν είναι σχετικό. Αν έχουμε τέτοιον ορισμό δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε στο μέλλον εκτός αν έχουμε παράρτημα. Δεν ξέρω αν η διαγραφή είναι η λύση. Ε, δεν ξέρω αν πρέπει να είμαστε κατά αυτού του ορισμού της σχετικής πληροφόρησης. Δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν ε, στιγμές όπου η σχετική ε, πληροφόρηση είναι κάτι το βασικό για να προσδιορίσουμε αν υπάρχει κατάχρηση. Θα συλλέξουμε τις ερωτήσεις, ή δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο. Κάινεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σχολιάσετε για τις προτάσεις σας και τις δικές σας παρεμβάσεις διότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Πώς θα σχολιάζετε λοιπόν τις προτάσεις σας. Οι προτάσεις σχετικά με το να δώσουμε περιτότερη αρμοδιότητα και ε, υπευθυνότητα στις ε, στους ε, παίκτες της αγοράς που ασχολούνται με την ανείχνευση. Θα ήθελα να δω και άλλοι πώς αντιδρούν σε αυτήν την πρόταση και πώς οι παίκτες της αγοράς θα μπορούσαν να δρουν με τρόπο πιο υπεύθυνο για να είναι το σύστημα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Τη δεύτερη ερώτηση είναι ότι η Κομισιόν έχει ε, τονίσει ορισμένες στρατηγικές του trading που θα πρέπει να ρυθμιστούν όταν έχουμε trading ε, μεγάλη συχνότητας. Αν θα υπάρχει γενική νομοθεσία και ίσως αργότερα αυτά να αναφερθούν ως παραδείγματα ή να έχουμε ειδική νομοθεσία η οποία να ε, ξεκαθαρίζει αυτές τις περιπτώσεις. Μήπως αυτές οι δυνητικές καταχρήσεις δεν θα μπορούσαν ε, να ε, θεωρηθούν ως καλά παραδείγματα και όχι ως πλήρης κατάλογος, εξαντλητικός κατάλογος. Και πώς θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε αυτήν την πρόταση με άλλους ε, τομείς του trading εκτός από το trading υψηλής συχνότητας. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ ενώπιον όχι λόγω της ζημιάς σε άλλους επενδυτές λοιπά αξίζει την προσοχή μας, αλλά κυρίως επειδή η εμπιστοσύνη των πολιτών στον χρηματοοικονομικό τομέα που ούτως ή άλλως έχει αποδυναμωθεί, με κάθε νέο σκάνδαλο εκ νέου αποδυναμώνεται και ε, γίνεται πιο ε, μικρών διαστάσεων. Η ζημιά που προκαλείται εδώ λόγω κατάχρησης θέσης αγοράς ε, στις συναλλαγές μπορεί να ποσοστοποιηθεί. Ξέρουμε ποιος είναι ο όγκος, ποιο είναι το μέγεθος αυτών των περιπτώσεων και των ζημιών και ποιοι πλήττονται. Δεύτερον, αυτή η ζημιά από την δημιουργία εναλλακτικών ε, δράσεων ή μορφών συναλλαγών παίρνει μεγαλύτερο όγκο και ακόμα περισσότερο επειδή ενδομεταξύ υπάρχουν δυνατότητες για το high frequency trading, συναλλαγές υψηλής συχνότητας, ταχύτατες δηλαδή σε μηδενικό χρόνο συναλλαγές. Και αυτό το οποίο αναφέρθηκε από την κυρία Χάρτμαν, είναι ρεαλιστικό να υποθέτει κανείς όταν έχουμε μια επισκόπηση και εποπτεία πρωτογενούς αγοράς, primary market surveillance, και υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα υπέρ αυτής της θέσης, ότι οι άλλοι συναλλασσόμενοι και φορείς είναι πρόθυμοι τα στοιχεία και τις πληροφορίες να τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους ώστε να υπάρχει το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα εποπτείας. Είναι ρεαλιστικό να υποθέτει κανείς με ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι κάτι θεωρητικό μόνο στην εξέτασή του. Τελευταίο σημείο. Είδαμε βλέπουμε ότι οι Εθνικέ Αρχέ εποπτείας έχουν διαφορετικές δυνατότητες. Σε κάποιες χώρες μπορούν μάλιστα και ως ένα είδο αστυνομίας να προβούν σε ποινικέ διώξεις. Σε άλλες χώρες μόνο διοικητικέ αρμοδιότητες έχουν και για την δίωξη ποινικά πρέπει να επιληφθούν του θέματος οι εθνικές αστυνομικές αρχές στη συνέχεια, οι, οι δικαστικές αρχές. Τι γίνεται λοιπόν εδώ, ερώτησή μου, ποιο ρόλο διαδραματίζουν, ποιο ρόλο θα έχει η ΕΣΜΑ μέσα σε αυτές τις διαφορές, σε αυτό το διαφορετικό πλαίσιο όσον αφορά τις αρμοδιότητες των εθνικών εποπτικών αρχών. Μπορεί ως καταλήτης να δράσει αυτή η αρχή στο μέλλον για την ΕΣΜΑ θα είναι πιο εύκολο κάτι τέτοιο ή θα δυσχεράνει το έργο της. Πώς μπορεί να καθοριστεί αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κέι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους σας για τη συμβολή σας σήμερα το απόγευμα. Την Παρασκευή ήμουν στο Παρίσι με μια ομάδα διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και διαθεσίμων που εκπροσωπούν Γάλλους επενδυτές όταν σχολίαζαν τα διάφορα θέματα σχετικά με την δομή της αγοράς και της καταχρήσης. Βεβαίως ασχολήθηκαν με το arbitrage trading ε, αλλά το κοινό του στοιχείο είναι ότι κινδυνεύουν να χάσουν το δάσος από τα δέντρα. Υπάρχει η μεταβλητότητα 10% μέσα στην ημέρα λόγω των φημών στην αγορά. Οι φήμες που κυκλοφορούν στην αγορά οδηγούν σε μεγάλη μεταβλητότητα και διακυμάνσεις στην αγορά. Είναι ένα θέμα τώρα που γίνεται σύνηθες αλλά έχουμε βεβαίως αυτή την μαζική κίνηση όταν υπάρχει μια ψεύτικη φήμη που κυκλοφορεί στην αγορά. Ίσως το πάνελ θα μπορούσε να σχολιάσει και τι μέτρα θα μπορούσαν να προταθούν για να ανταπιτοπιστούν αυτές οι ψευδοφήμες που κυκλοφορούν. Ευχαριστώ από τους πράσινους. Μίγκουαλ Ποτέσου, θέλει να σχολιάσεις. Όχι, δεν είναι εδώ. Όλα. Είναι η σειρά σου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, παρέμβαση. Ε, Σύρπα και Βόλφ έχουν θέσει τις ερωτήσεις που ήθελα και εγώ να θέσω. Αλλά σχετικά με την αξιολόγηση αντικτύπου, αν ε, δούμε αυτό το έγγραφο, δεν είναι τόσο σαφές ότι υπήρξε αύξηση ε, συμπεριφορών κατάχρησης αγοράς. Και αυτό σχετίζεται με την ερώτηση του κυρίου Κλίντς επίσης. Διότι γνωρίζουμε πράγματι ότι υπήρξε τρομερή αύξηση σε τέτοιες περιπτώσεις σύμφωνα με τις στατιστικές εδώ στην αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν. Αυτή δεν είναι η περίπτωση. Θα ήθελα τα σχόλιά σας σχετικά με το θέμα αυτό στην χειραγώγηση αγοράς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ερώτηση για τον εισηγητή. Στην, στον κανονισμό λέει ότι δίνει ή θα μπορούσε ε, να δώσει απατηλά ε, σημάδια ε, για τα, τις κυρώσεις της ποινικέ σχετικά με την χειραγώγηση ότι δίνει ε, ψευδή στοιχεία ή απατηλά στοιχεία. Εσείς είστε οι εμπειρογνώμονες. Πώς ερμηνεύετε αυτό, αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπαν οι προηγούμενοι για να υπάρχει φυσικά κάτι το ποινικό πρέπει να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Αυτό είναι σαφές. Θέλουμε λοιπόν εμείς να προωθήσουμε την εμπιστοσύνη στις αγορές. Αυτό είναι το βασικό. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ αυτής της διαδικασίας ότι θα πρέπει η νομοθεσία, οι νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι ιδιαίτερα αυστηρές. αλλά αν είναι να διστάζει κανείς, είναι προτιμότερο νομίζω να προχωρήσει. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση βρισκόμαστε σε ένα πεδίο πραγματικά με ουσιαστικές ελλείψεις γνώσεων σχετικά με τους τρόπους ανείχνευσης κάποιων καταχρήσεων των αγορών. Αν κυκλοφορεί κανείς στο City ακούει πάρα πολλές φήμες, ακούει πάρα πολλές υποψίες να ανταλλάσσονται στους διαδρόμους και εγώ εδώ ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους μου, τους φιλελευθέρους, αυτό το οποίο λέω ίσως να μην είναι πολύ φιλελεύθερο, αλλά είναι σαφές ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, τουλάχιστον τις περισσότερες περιπτώσεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι επιθετική εδώ, θέλω να είμαι απαιτητική εφόσον, α, α, να μην, εφόσον δεν δημιουργούμε βέβαια καταστάσεις όπου στην ουσία ανοίγουμε παγίδες στις οποίες κινδυνεύουμε εμείς οι ίδιοι να πιαστούμε. Σχετικά με την κατανομή και την κυκλοφορία των πληροφοριών υπάρχουν διάφορα θέματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα ανταλλάσσονται οι πληροφορίες και το επίπεδό τους και το επίπεδο λεπτομέρειας και πόσο εύκολο είναι να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά όλες τις πλευρές της νομοθετικής δραστηριότητας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να βελτιώσουμε την εποπτεία σε πραγματικό χρόνο, τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. εφόσον γίνεται φυσικά αυτό χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις και χωρίς να φύγονται κάποιοι περισσότερο από κάποιους άλλους. Αυτά ήθελα να κάνω σαν σχόλια, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από πλευρά των μελών του Κοινοβουλίου. Ίσως εδώ θα πρέπει να ζητήσω τις απόψεις αυτών που πήραν το λόγο προηγουμένως ανάποδα. Προσπαθήστε παρακαλώ να μην ξεπεράσετε σε ένα-δυο λεπτά ο καθένας. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο δυστυχώς. Ε, σύντομος θα είμαι. Σχετικά με τις πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να καταγράφονται ακόμα και όταν δεν είναι επεξεργασμένες η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι πληροφορίες που είναι στη διάθεσή μας ε, δεν ε, είναι επεξεργασμένες και φυσικά ε, με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές δεν είναι κυκλοφορήσιμες. Ξέρουμε ότι πολλές περιπτώσεις M&A έχουν ξεκινήσει από απλές συζητήσεις ανάμεσα σε υπευθύνους επιχειρήσεων και είναι σαφές ότι τέτοιου είδους στοιχεία και τέτοιου είδους ίχνη θα έλεγα δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν εκτός και αν κάθε επιχείρηση θεωρεί ότι οφείλει να το κάνει αυτό στα πλαίσια της σωστής της ενημέρωσης. Το θέμα δεν είναι για την ανταλλαγή των δεδομένων μόνο τεχνικό υπάρχουν θέματα που αφορούν όχι μόνο αυστηρά την συναλλαγή, αλλά υπάρχουν και στοιχεία των πελατών, σαν παράδειγμα, και εκεί υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με την δυνατότητα κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών. Βέβαια πολλές φορές τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει σε επίπεδο συναλλαγών και σε επίπεδο έκδοσης εντολών. ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου υπάρχουν καταχρήσεις σε πολλές ταυτόχρονα αγορές. Οι καταχρηστικές πρακτικές, έχει τεθεί το θέμα, αν θα πρέπει να είναι στο πρώτο επίπεδο του κανονισμού ή αν θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ δυνατότητα έτσι ώστε να ορίσουμε ορισμένες έννοιες μέσω τεχνικών standards. Όπως είδαμε με την οδηγία για τις αγορές, υπάρχει μια σαφή συζήτηση για κατευθυντήριες γραμμές ερμηνείας συγκεκριμένων καταστάσεων και σε σχέση με το insider information και σε σχέση με τις καταχρήσεις των αγορών. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης, μιας δυναμικής βελτίωσης του τρόπου εποπτείας των αγορών, έτσι ώστε να προσαρμοστούν οι περιγραφές των συγκεκριμένων συμβάντων στην πραγματικότητα των αγορών σχετικά τώρα με τις διαφορετικές αρχές από τις διαφορετικές χώρες και σε ποιο βαθμό αυτό δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της ΕΣΜΑ, σαν παράδειγμα. Όχι. Η εναρμόνιση την οποία άλλωστε ε, οδηγεί, εισάγει η πρόταση αυτή θα καταστήσει τη συνεργασία ανάμεσά μας και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ε, μιλάω σαν έσμα, ακόμα καλύτερα έτσι και αλλιώ η ΕΣΜΑ είναι προϊόν, αν θέλετε, της συνεργασίας ανάμεσα στις εθνικές αρχές. Είναι κάτι το οποίο δουλεύει. Για το αν υπάρχουν αυξήσεις στον τομέα των καταχρήσεων των αγορών. Εγώ εδώ θα ήθελα να ήμουν επιφυλακτικός σε σχέση με, με φήμες, ε, ε, με ελέγχους τιμών σε καθημερινή βάση κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό για την εικόνα που ισχύει σήμερα. Κάπου κάπου μπορεί να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις, αλλά όχι όμως σε μόνιμη βάση. Το θέμα είναι δεν γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων αν υπάρχει μια παράνομη μορφή επικοινωνίας ανάμεσα σε εμπλεκομένους στις αγορές που δεν θα έπρεπε να υπάρχει θα πρέπει να υπάρχουν εξισιοδοτήσεις σε σχέση με τη συγκέντρωση των στοιχείων που να οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων περίπου αυτόματα. Αυτό δεν ισχύει ιδιαίτερα για το insider dealing, ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε ε, τα δεδομένα που έχουμε σήμερα με τα δεδομένα του 8, 9 και 10. Το επίπεδο εποπτείας δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ και γι' αυτό δεν πρέπει να καταλήγουμε σε βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπιστία της αγοράς, η οποία υποτίθεται είναι λιγότερο αξιόπιστη από ό,τι 5, 6, 10 χρόνια πριν. Πρέπει να επιτεχύνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Θα επικεντρωθώ στα θέματα που αφορούν την κοινή χρήση τέτοιων στατιστικών στοιχείων, αν έχουμε τέτοια στοιχεία για την κατάχρηση αγορών ή όχι λόγω του κατακαιρματισμού των αγορών. Αυτό ζητήθηκε και κατά το παρελθόν από εμάς. Από τότε, μια και δεν έχουν εντολή πρόσβαση οι συναλλασσόμενοι στις αγορές των άλλων, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η εμβέλεια, αν δηλαδή η συχνότητα αυτή έχει αυξηθεί ή όχι στην κατάξη αγορών. Το μόνο που μπορούμε να δούμε φυσικά είναι ότι είναι κατακαιρματισμένη η αγορά. Είναι πολύ πιο εύκολο να τεθούν οι εντολές και οι παραγγελίες σε διάφορα πλατό, ε, σε, διάφορα, ε, σε διάφορες πλατφόρμες και είναι δύσκολο το έργο της εποπτείας. Και έχουμε και κάποιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για χειραγώγηση αγορών που πάντα συμπεριλαμβάνουν δύο ή τρεις διαφορετικές έδρες ως ε, γήπεδα εντός εισαγωγικών. Φυσικά αν γίνεται ταυτόχρονα σε διαφορετικά γήπεδα είναι ευκολότερο να μην ανοιχνευτεί κάτι. Όμως ε, ε, έχοντας την κοινή αυτή εποπτεία θα είμαστε πραγματικά ανήσυχοι αν δεν ελαμβάνονται μέτρα και διαβήματα κατά της κατάστασης αυτής. Θα ήταν πολύ αρνητικό για την ευρωπαϊκή αγορά αν ξεσπούσε ένα σκάνδαλο λόγω της κατάχρησης αγορών και διαπιστωνόταν ότι συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση επί χρόνια και ήταν τόσο εύκολο να γίνεται επειδή είναι κατακαιρματισμένες οι αγορές και είναι εύκολο τέτοιου είδους κέρδος. Θα μας ανησυχούσε ιδιαίτερα. Μας ανησυχεί πράγματι και πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε. Τώρα, το να συμμεριζόμαστε στοιχεία με άλλους, μια και είμαστε μια εποπτική αρχή με εποπτικές αρμοδιότητες, ε, από πλευράς νομοθεσίας και της άδεια μας πρέπει να διαφοροποιούμαστε από τις εμπορικές μας συναλλαγές και δράσεις. Είμαστε λοιπόν ανεξάρτητοι ως όργανο και υπό μια άδεια υπό την οποία δρούμε, δραστηριοποιούμεθα. Έχουμε αυτού του είδους την εμβέλεια και δεν θα ε, υπήρχε δυνατότητα ή άλλο περιθώριο, μια και από πλευρά νομοθεσία δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι δυνατότητε για άλλου σκοπού. Αυτό έχει συζητηθεί και ε, με άλλου και όλοι συμφωνούν φυσικά ότι κάτι πρέπει να γίνει από πλευρά μα. Να καταπολεμηθεί η κατάσταση κατάχρηση ε, των αγορών. Το καλύτερο είναι πρωτογενώ να δράσουμε στην πρωτογενή αγορά να έχουμε συνολικά τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ίσως για να πάμε ανάποδα για να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε. Η ιδέα ότι υπήρχε λέει δραματική αύξηση στην κατάχρηση αγορών είναι μάλλον εσφαλμένη. Η κατάσταση είναι ότι ξεκινήσαμε να εξετάζουμε και να ρυθμίζουμε τις αγορές με πιο όριμο τρόπο. Και γι' αυτό ανακαλύψαμε ότι οι περιπτώσεις κατάχρησης αγορών μπορεί να υφίσταται σε κάποια υπολείμματα ή κατάλοιπα. Πρέπει να κατανοήσουμε όμως ότι οι συναλλαγές ε, είναι σαν ένα ένα Έχει τις καλές στιγμές της, έχει τις αρνητικές στιγμές της. Είναι ένα σενάριο υποεξέλιξη. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ρυθμίζουμε με στόχο να ρυθμίζεται η αγορά με καλό, εύθετο τρόπο, αντί να υιοθετούμε κάποιες ε, τεχνολογικές ε, εξελίξεις, γιατί έτσι θα ήταν δύσκολο να σημειωθεί πρόοδος διότι σε σχέση με τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας βρίσκονται υποεξέλιξη δημιουργούν πολλές ομάδες, ε, υποομάδες ε, υψηλής συχνότητας ε, συναλλαγών και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς αυτή την συνιστόσα. Στο τέλος τέλος, ενώ θέλουμε να εκριζώσουμε τις κακές αρνητικές πρακτικές, πρέπει να το κάνουμε σε μια συνολική, σε ένα συνολικό πεδίο και επίπεδο για όλους τους εμπλεκόμενους, για την ευμεταβλητότητα, για τη μεταβλητότητα. Δεν νομίζω ότι οι φήμες είναι εκείνες που δίνουν έναυσμα είναι σαν σπίθα η φήμη, ο ψήθυρος. Αν πέσει ε, σε, προσά, σε ε, ξερά χόρτα ανάβει αμέσως ε, φωτιά από αυτή τη σπίθα. Και υπάρχουν εδώ ένας ε, μια ολόκληρη πληθώρα μακροοικονομικών ε, συνιστοσών και παραγόντων και όχι μόνο κάποια φήμη ψήθυρος που προκαλούν τη ζημιά στο τέλος ε, ή για την παράνοια της αντίδρασης που σημειώνεται από πλευράς του λογισμικού. Και σε σχέση με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές αυτά έχουν ζωτική σημασία πρέπει να πω, διότι οι εθνικοί ρυθμιστές μπορεί να υπερρυθμίζουν τα πράγματα και σε αυτό τον, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στραγγαλίζουν την ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων και στοιχείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα μπορεί να ήταν εποφελές εγχείρημα. Για την πρώτη ερώτηση τώρα στη συνέχεια της κυρίας Μακάρθη. Θα έλεγα ότι μια αποτελεσματική εφαρμογή του 6A, δηλαδή η παραδοσιακή έννοια και ορισμός του της ε, ενδοπληροφόρησης, καθώς επίσης η εμπλοκή των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων θα ήταν επαρκές στοιχείο για να κατανοήσει κανείς και να αποφύγει τα προβλήματα τα οποία τίθενται σε σχέση με την ΕΣΜΑ. Υπάρχει κάποια πληροφορία που δεν μπορεί να τύχει χρήση Όμως αυτό εκ πρέπει να ισχύει σε σχέση με τα αποκαλυπτόμενα στοιχεία των, ε, της ενδοπληροφόρησης. Πρέπει να δίνονται περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες και να αποσαφηνίζεται σε σχέση με τα στοιχεία τι αποκαλύφθηκε και τι όχι για την επίλυση των αμφισημιών και προβλημάτων και για την αντιμετώπιση της ανάγκης να υπάρξει ένας νέος κανονισμός. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ με την υποκατάσταση της πρώην οδηγίας ε, ενισχύει με ένα νέο κανονισμό. Όμως ουσιαστικά πιστεύω ότι και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει μια μελέτη που να αποσαφηνίζει τι συνέβη σε πολλά κράτη-μέλη. Αν σε πολλά κράτη-μέλη είτε ρητά ε, όπως στην Ισπανία είτε έμεσα όπως στην Ιταλία είτε στη, όπως στη Γαλλία με τον κανονισμό EMF είτε σε σχέση με τη Γερμανία είτε δεν προσαρμόζονται, δεν συμμορφώνονται σε σχέση με τις ε, διαδικασίες και κανονισμούς ε, αντιμετώπισης κατάχρησης στην αγορά, ε, είτε δεν, για την αντιμετώπιση της ενδοπληροφόρησης, αυτά θα πρέπει να μας κάνουν να προβληματιστούμε για να κατανοήσουμε καλύτερα ότι χρειάζεται στενότερη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών σημαντικότερος και ισχυρότερος ρόλος της ΕΣΜΑ μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής και των, της δικαιοδοσίας της. Όμως Πρέπει να το δούμε αυτό και έτσι το 6ε θα έπρεπε να διαγραφεί και να χρησιμοποιείται πιο, ε, πιο αποτελεσματικά το 6α. Ευχαριστώ. Σχετικά με το πρώτο θέμα για την ε, κανονισμό για το, το trading υψηλής συχνότητας, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ειδικό κανονισμός για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι οι τέσσερις διαγνωστικές σημαίες νομίζω ότι ε, μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν. Ε, διάβασα τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΣΜΑ. Νομίζω ότι αυτές είναι ένα καλό πλαίσιο σχετικά με την ιδέα να βασιστούμε πολύ περισσότερο σε εποπτεία από επενδυτικές εταιρείες. Υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα διότι ε, το trading υψηλής ε, συχνότητας ε, γίνεται μια υπηρεσία με ειδική άδεια στην MIFID 2. Όταν λοιπόν κάποιος έχει την άδεια, έχει το διαβατήριο, θα πρέπει να μπορεί εσωτερικά να εποπτεύει αυτήν την υπηρεσία. Αν υπάρχει περισσότερα περιπτώσεις κατάχρησης δεν ξέρω ε, κάθε χρόνο έχουμε ε, περίπου τον ίδιο αριθμό, 15. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρομερή αύξηση και σχετικά ε, με την, της σύνδεση ανάμεσα στις φήμες και το trading υψηλής συχνότητας. Μπορεί αυτό να είναι η βάση της κατάχρησης αν υπάρχει ε, μια φήμη αυτή ε, κυκλοφορεί από έναν trader ε, και, που, και έτσι επηρεάζεται η τιμή και αυτό αυξάνει την κίνηση υπέρ του προϊόντος, διευρύνει την όλη κίνηση. Δεν έχουμε όμως σαφή εξήγηση για τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με το άρθρο 6.1 ε, βεβαίως ε, συμφωνώ πλήρως ότι η εσωτερική πληροφόρηση οδηγεί σε κατάχρηση. Υπάρχει επίσης μια ανάγκη να πούμε τι είναι κατάχρηση. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, πληροφορίες που αν χρησιμοποιηθούν δεν οδηγούν σε κατάχρηση. Γι' αυτό αν έχουμε την, τις σχετικές πληροφορίες πρέπει να μπορούμε να δούμε αν είναι χρήσιμες, αν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι αποτυχία να πληρούνται τα πρότυπα και οι κανόνες. Ε, η κυρία Πιετικά ε, ρώτησε για εποπτεία σε πραγματικό χρόνο, επίσης ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών για MTF. Ναι, η εποπτεία της αγοράς δεν είναι επαρκής. Έχουμε τον κατακαιρματισμό από την MIFID 1 και θα πρέπει να έχουμε εποπτεία της αγοράς σημαντική. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά νομίζω, νομίζω ότι η ΕΣΜΑ ασχολήθηκε και ότι ε, έχουν την πραγματογνωμοσύνη, την ανεξαρτησία που απαιτείται για να ε, εξασφαλίσουν εμπιστοσύνη και νομίζω ότι όταν υπάρχουν ε, για τα στοιχεία διαμάχες ανάμεσα στις ε, τράπεζες έχει σημαντικό ρόλο να πέσει. Επίσης ε, ρωτήσατε για τις στρατηγικές υψηλής συχνότητας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προσδιοριστούν ειδικά στον κανονισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα εργασίας που να τις εξετάζει. Ε, μπορεί να υπάρχει αταξία στην αγορά, όχι η κατάχρηση, μπορεί να υπάρχουν θέματα εμπιστοσύνης, μπορεί να υπάρχουν αδυναμίες τεχνολογίας όπως προσδιορίσε η ΕΣΜΑ. Επίσης ε, ρωτήσατε ε, για την ποσοτικοποίηση. Νομίζω ότι όταν αναφέρθηκε αυτό προηγουμένως εξεπλάγει. Νομίζω ότι η κυρία Σουίμπερ μίλησε για το θέμα αυτό. Ε, στην αγορά, οι ψεύτικες φήμες έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να διερευνήσουμε τις περιπτώσεις αυτές, να παρακολουθήσουμε τι έχει γίνει. Ο Χερ Σμιτ ανέφερε σε ορισμούς για την χειραγώγηση. Υπάρχουν διαφορές στους ορισμούς, υπάρχουν ορισμένα τεχνικά θέματα ε, θα πρέπει ε, έχουμε από τη μια πλευρά τους τίτλους, τα χρεόγραφα και από την άλλη πλευρά επενδυτικά προϊόντα. Επίσης το θέμα της πρόθεσης ε, την πρόθεση, αν υπάρχει πρόθεση, θα πρέπει να ερευνήσουμε τις περιπτώσεις, αν είναι κατάχρηση, αν έχουμε πραγματική αξία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χρήση ε, των πληροφοριών πρέπει να απαγορευτεί, όχι η κατοχή πληροφοριών, ε, διότι υπάρχει κατοχή σε περιπτώσεις όπου μπορεί κανείς να υποθέσει ότι υπάρχει ενοχή, ενώ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της ακρόασης. Δίνω τον λόγο στον εισηγητή για μερικές παρατηρήσεις για το κλείσιμο. Στην εισηγήτρια θα είμαι σύντομη για να τηρήσουμε το χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που μοιραστήκαν τις γνώσεις τους μαζί μας. Τις προτάσεις σας θα τις λάβουμε υπόψη, θα τις εξετάσουμε με τους σκιώδεις εισηγητές και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να διαρωτηθούμε αν υπάρχει αύξηση στις περιπτώσεις κατάχρησης είχαμε μια, ήδη μια οδηγία για το θέμα των καταχρήσεων. Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να έχουμε αύξηση στις περιπτώσεις καταχρήσεων. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχουν ευξημένες ευκαιρίες και δυνατότητες για καταχρήσεις. Έχουν πολλαπλασιαστεί ε, τα σημεία για το trading, για τις ε, συναλλαγές σε 7 διαφορετικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αύξηση των ετοιμάτων για, ε, ε, για στοιχεία από 500 σε 600. Δεν σημαίνει ότι υπήρξε αύξηση καταχρήσεων, αλλά θα πρέπει η νομοθεσία την οποία επεξεργαζόμαστε να προτρέξει, να μπορέσει να προλάβει ορισμένες καταχρήσεις. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους σκιώδεις συγητές. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την πρόταση εν ευθέτω χρόνο, ούτως ώστε να εξεταστεί από την Επιτροπή. Ευχαριστώ για αυτούς που ενδιαφέρονται. Θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή στις 6 Φεβρουαρίου μετά την παρουσίαση ενός σχεδίου έκθεσης στις 26 Μαρτίου και προθεσμία στις 24 ε, Απριλίου για τις ε, τροπολογίες και να εξεταστούν ε, στις 30 Μαΐου στις Επιτροπής και στις 18 Ιουνίου αν χρειαστεί και ψηφοφορία στις 9 Ιουλίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό αν έχουμε βεβαίως περισσότερες τροπολογίες από ό,τι αναμένεται, αυτό βεβαίως θα έχει επιπτώσει. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Το επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία, αλλά ε, θα, αφήσουμε, ε, θα διακόψουμε για μερικά λεπτά, ούτως ώστε όσοι θέλουν να φύγουν να μπορέσουν να φύγουν. Ευχαριστώ τα μέλη του πάνελ. Can you take your seats? I think... Παρακαλώ καθίστε, είμαστε αρκετοί τώρα και μπορούμε να συνεχίσουμε. Jolly well. A letter that we might. Καθίστε παρακαλώ. Καθίστε για να προχωρήσουμε με τις ε, ψηφοφορίες πιο αποτελεσματικά. Προχωρούμε τώρα και θα ψηφίσουμε την έκθεση του Ζαν Paul για τις εισφορές συνεισφορά στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης. Θα αναμείνω μέχρι ότου καθίσει ο εισηγητής στο κάθισμά του, στο εδρανό του. Εντάξει, Καταφέρνουμε να είμαστε σχεδόν με το χρονοδιάγραμμα στην ώρα μας. Καλά, καλά προχωρήσαμε, καλή δουλειά. Όλοι έτοιμοι λοιπόν για τις ψηφοφορίες. Έτοιμοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Αρχικό κείμενο τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 11. Α, μια κάρτα λείπει σε κάποιο μέλος. Λοιπόν, Άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει λοιπόν, ψηφίσατε όλες και όλοι. 38 έχουν την, είναι που έχουν δικαίωμα ψήφου, 37 ψηφίζουν, κάποιος απέχει. Τέλος πάντων λίγη ψηφοφορία. Αποτέλεσμα 18 υπέρ, 17 εναντίον και μία ακόμα η Σιλβή 19 λοιπόν υπέρ εγκρίθηκε επανερχόμαστε λοιπόν σε 19-18 πάλι με μία ψηφοδιαφορά εγκρίνεται, εγκρίνεται. εντάξει Φιλίππε. τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 13 θα ελέγξουμε λοιπόν θα ψηφίσουμε, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία τοπολογία 12. Μια άλλη κάρτα που λείπει, απουσιάζει, αναφέρεται. Εντάξει λοιπόν, ψήφισαν όλοι. Τρεις είναι που δεν ψηφίζουν, δεν συμμετέχουν. Ένας τώρα που δεν ψηφίζει. Εν πάση περιπτώσει, λίγη ψηφοφορία τώρα. Και το αποτέλεσμα απερίφθη σαφώς, ε, όπως είχα προείπει. Τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός Β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Γ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Αρχικό κείμενο τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 26, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 27, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Αρχικό κείμενο, στο σημείο 4 υπέρ κατά, στην παράγραφο 5 εγκρίθηκε, τροπολογία 28 υπέρ κατά, αποχές εγκρίθηκε, Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός ε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός σίγμα τάφ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 39 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε προφορική τροποποίηση από την, τους σοσιαλδημοκράτες κάπου. Εντάξει, η προφορική τροποποίηση για την τροπολογία 40. Υπέρ λοιπόν, κατά. Δεν συμμετέχετε. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επ' αυτής. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι η προφορική τροποποίηση των σοσιαλδημοκρατών. στην παράγραφο που έχει 6α μετά και είναι αντί της τροπολογίας 40 ψηφίσαν όλοι κάποιοι άλλοι ακόμα πρέπει να συμμετάσχουν δύο ακόμα που πρέπει να ψηφίσουν λίγη τώρα η ψηφοφορία σε λίγο πέρας λοιπόν ψηφοφορίας και αποτέλεσμα συντριπτικά εγκρίθηκε <clears throat> παρότι δεν είχαμε πολλούς να συμμετέχουν με ανάταση χειρών τώρα τροπολογία 41 για, σε σχέση με τον εισηγητή σε δύο τμήματα Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Σε τμήματα ψηφοφορία για την προφορική όχι, όχι, όχι για την προφορική τροποποίηση, αλλά σε τμήματα επί της ίδιας της τροπολογίας. Λοιπόν, όσοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 41, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία. Θα το ελέγξουμε αν θέλετε. Δεύτερο τμήμα της 41. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και πιο πολύ τώρα εδώ από ό,τι βλέπω. Απορρίφθηκε λοιπόν. 18 υπέρ, 20 εναντίον. Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα της 41. Ο κύριος Φακμακ θα έλεγα έχει τη δική το είναι όμω υπέρ 19 έναντι 20 παρόλα αυτά απορρίπτεται πάλι 20-19 ναι ναι έχετε βάλει την κάρτα σα απορρίπτεται παρόλα αυτά με μια ψήφο διαφορά όχι δύο εν πάση περιπτώσει λοιπόν τροπολογία 42 υπέρ κατά άποχες θα έλεγα εγκρίνεται συμβιβασμό ζ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός ΙΤΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 53 τροπολογία ως προσθήκη στο συμβιβασμό υπέρ κατά Τροπολογία 53 βέβαια. Λέει εδώ μπορεί να ψηφιστεί ως προσθήκη στο συμβιβασμό ΙΤΑ. Εντάξει. Τροπολογία 53. Εισηγητά τι λέτε. Το παρακολουθείτε. Είσαστε σύμφωνος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και πάμε τώρα στον συμβιβασμό ΙΤΑ Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμ... Ε, τροπολογία 62. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τοπολογία 64 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίθηκε. Συμβασμός ε, ΙΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 69 τροπολογία υπέρ κατά αποχές είναι πολύ στενό το αποτέλεσμα. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Και μία προσθήκη ακόμα επιπλέον, 21 εναντίον τώρα με 19 υπέρ. Έτσι λοιπόν καταψηφίζεται. Η τροπολογία 70 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίθηκε. <clears throat> Συμβιβασμός L υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίθηκε. Η 77 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός N μια, μια στιγμή σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές και αυτό το δεύτερο εγκρίθηκε. Τροπολογία 81 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός N υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός O υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Υποκεφάλαια 2 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός π υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τοπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Αρχικό κείμενο, παράγραφο 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Παράγραφος 16, τροπολογία 96, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 97, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 98, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Αρχικό κείμενο τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 99, υπέρ, κατά, αποχές, Δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 99 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα με 19 υπέρ 21 εναντίον. απορρίφθηκε όμως. Αρχικό κείμενο τώρα, παράγραφος 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Q υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τοπολογία 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Αρχικό κείμενο τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε αρχικό κείμενο τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 109 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 109 ψηφίζουμε άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία παρακαλώ ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας τώρα και αποτέλεσμα τέλος λίγη ψηφοφορία και απορρίφθηκε 18 υπέρ 24 τώρα εναντίον κιόλας αρχικό κείμενο τώρα παράγραφος 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε παράγραφος 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τροπολογία 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Παράγραφος, 100, ε, συγγνώμη, παράγραφος 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 111 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 1 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. <coughs> Αιτιολογική σκέψη 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Αιτιολογική σκέψη σκεπτικό 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Σκεπτικό 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Αιτιολογική σκέψη στο, στην τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε την τελική ψηφοφορία στο κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Δύο ακόμα που λείπουν για να ολοκληρωθεί ο αριθμός. Συνεχίστε να ψηφίζετε. Εντάξει, τέλος ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα 35 τώρα πλέον υπέρ, Τρεις εναντίον, τέσσερις αποχές. Εγκρίθηκε συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Okay. Are we ready for the next If you could take your seats, please. καθίστε και να προχωρήσουμε στο σημείο 16. Administrative cooperation in the... Διοικητική συνεργασία στο θέμα των ειδικών φόρων. Please, conversations outside. It's still conversations outside, please. Λοιπόν, καθίστε. Γκέι Μίτσελ, θα μιλήσει εξ ονόματος ε, του εισηγητή, του κυρίου Κάζα. Δυστυχώς, λόγω απρόβλεπτων υποχρεώσεων, ο κύριος Κάζα δεν είναι δυνατό να είναι μαζί μα σήμερα, μου ζήτησε όμως να παρουσιάσω την έκθεσή του. Και θα ενημερώσω και τον κύριο Κάσα για τις συζητήσεις που πιθανώς να ακολουθήσουν βάση είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού του 2004 που δημιούργησε ένα νομικό πλαίσιο για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να ενημερωθεί έτσι ώστε να παράσχει τη νομική βάση για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι η εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του CMCS των ειδικών φόρων. Έχει σαν επιπλέον στόχο την εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών έτσι ώστε η ανταλλαγή πληροφοριών να είναι πιο αποτελεσματική σε επίπεδο ταχύτητας και αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή σε εφαρμοστεί πλήρως ένα τέτοιο σύστημα θα είναι καθοριστικό στη μείωση των απατών. Το σύστημα θα μειώσει επίσης και τα διοικητικά άχθη από πλευράς των αρμοδίων αρχών στα πλαίσια της ανάγκης αμοιβαίας συλλογής ε, πληροφοριών η οποία θα μειωθεί. Θα μειωθούν επιπλέον διοικητικά βάρη επίσης και για τις ε, επιχειρήσεις μέσω της συστηματικής συλλογής πληροφοριών. Ο κύριος Κάζα υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρεί ότι τα μέτρα τα οποία έχουν σαν στόχο την απλοποίηση των διαδικαστιών από πλευράς κρατών μελών και επιχειρήσεων είναι καλοδεχούμενα. Ένα ταχύ και αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών είναι θεμελιώδες έτσι ώστε να καταστήσει ικανές τις αρμόδιες αρχές να καταπολεμήσουν την απάτη. Ο αναθεωρισμένος κανονισμός θα βελτιώσει την ανείχνευση και την ακολουθούμενη μείωση των διαδικασιών απατών κτλ. Γίνονται ορισμένε προτάσεις τροπολόγησης ε, των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες τροπολογίες έχουν στόχο να διευκρινίσουν καλύτερα το κείμενο της Επιτροπής, το 4. Στα πλαίσια των πληροφοριών από τα κράτη-μέλη, ο ρόλος της Επιτροπής δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην περίληψη αλλά και στην ανάλυση των στοιχείων αυτών. Η τροπολογία 5 αλλάζει τη χρονική περίοδο αναθεώρησης από τα 5 στα 3 χρόνια. Ο κύριος Κάσα θεωρεί ότι τα 3 χρόνια είναι προτιμότερο και περιμένει και την ιδέες των συναδέλφων γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Μπούλμαν, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε Μίτσερ και ευχαριστώ και τον συνάδελφο Κάζα φυσικά για το ότι έκαναν αυτοί, ανέλαβαν αυτό το έργο. Για τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα μπορώ να πω ότι χωρίς επιφυλάξεις υποστηρίζουμε αυτό το έργο. Πρέπει το σύστημα να γίνει ταχύτερο, να εξυγχρονιστεί οπωσδήποτε και πρέπει στις τεχνικές λεπτομέρειες να συνεχίσουμε το έργο μας ώστε η υποστήριξη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές αυτών των στοιχείων να υποστηριχθεί. Όλα αυτά βοηθούν. Ό,τι βοηθά να αποφύγουμε φοροδιαφυγή και φοροαπάτη. Ό,τι βοηθά η κάλυψη φορολογική να γίνεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο και η βάση δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών να ενισχυθεί. Θα τύχει της πλήρους υποστήριξής μας και γι' αυτό πιστεύω ότι στο τέλος τέλος πολύ γοργά θα καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Philippe. oh, hang Δεν είσαστε στον κατάλογο. Δεν το είχα σημειώσει τον σκιώδη της Άλντε των Φιλελευθέρων. Παρ' όλα αυτά έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Πρώτο εσεί Πρώτος εσείς λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ούτως ή άλλως πριν από 15 λεπτά με διόρισαν να παρέμβω. Από κοινού με τον κύριο Κάζα είχαμε παρακολουθήσει αυτό το έργο και προηγούμενα και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και παρότι είναι πολύ, πολύ τεχνικό και περίπλοκο ζήτημα, είναι θεμελιώδου σημασία, ζωτική σημασία να σημειωθεί πρόοδο. Να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε για αυτή τη συνεργασία στην Ευρώπη. Τώρα, γενικά είμαι λοιπόν υπέρ. Υπέρ τη πρόταση που προέρχεται από τον κύριο Κάζα Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας λοιπόν για να καταλήξουμε σε μια πιο αποτελεσματική και ταχύτερη διοικητική διεκπαιρέωση που θα μειώσει ουσιαστικά τη γραφειοκρατική επιβάρυνση, το γραφειοκρατικό βάρος. Τώρα, σε σχέση με την τεχνική ουσία αυτής της πρότασης, κάποια λίγα σχόλια ακούστηκαν. Δεν ξέρω, εσείς κύριε Μίτσελ θα μπορούσατε να απαντήσετε έγκριση σε σχέση με το προτινόμενο άρθρο 15 σημείο εδάφιο 4 όπου καθορίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή σε ποιες περιπτώσεις οι εθνικές αρχές ε, τέτοια συστήματα ε, ε, ηλεκτρονικούς υπολογισμούς, υπολογιστές θα τα θεωρούσαν μη προσπελάσιμα. Χρειάζονται αποσαφηνήσεις εδώ. Δεν είναι σαφές τι θέλει επίσης να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το άρθρο 19 θα έπρεπε σαφώς να λέγεται ότι η διεύθυνση στο Μητρό SED θα πρέπει να είναι η ίδια όσον αφορά τα στοιχεία σε σχέση με εκείνον που είναι αποδέκτης των αγαθών όσον αφορά τις σχετικές διατάξεις. Θα μπορούσε έτσι λοιπόν να ρυθμιστεί το θέμα. Μία πρόταση είναι στο άρθρο 9 εδάφιο 2 να προσθεθεί μία αναφορά για ποια διεύθυνση θα προτιμούσε ο αποδέκτης, ο αποδέκτης των αγαθών αναφέρεται όσον αφορά τη χώρα του. Επίσης, σε σχέση με την έγκριση του Μητρώου SED, σε σχέση με το άρθρο 9.2, που θα μπορούσε να είναι η επιβάρυνση για κάποιες εθνικές αρχές, θα έπρεπε να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι μόνο εφάπαξ ε, κόστος και διαδικασία θα έπρεπε ε, να λαμβάνεται υπόψη να ολοκληρώσω. Θα πρέπει να είμαστε ίσως πιο τολμηροί, κάπως πιο τολμηροί από πλευρά της δικής μας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Είναι αδύνατο, είναι ανέφικτο να σκεφτεί κανείς ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε καν κύριε Μίτσελ όπως ε, μια κοινή αρχή για το ΦΠΑ, ΦΠΑ όσον αφορά το κοινό πακέτο φορολογικών μέτρων αυτό τι είναι, αυταπάτη, χήμερα ή θα μπορούσε να, να εφαρμοστεί. Διότι πολλά περισσότερα θα μπορούσαμε να κάνουμε σε σχέση με το ΦΠΑ, να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και την ε, παράκαμψη ε, καταβολής των φόρων, ώστε να, να αποτελεί αυτό ένα τμήμα της καλώς λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Φιλίπ, ε, κάποια μέρα θα έπρεπε να γίνομαι σύντροφοι, δεν ξέρω. Όχι, όχι, αναφέρομαι στα όσα είπες. Είναι ίσως μια προοπτική που πρέπει να λάβουμε υπόψη, δηλαδή να έχουμε μια αρχή για τον ΦΠΑ ευρωπαϊκή και μέσα στο πνεύμα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Και νομίζω ότι αξίζει να μπει σε μια αιτιολογική σκέψη αυτό. Συμφωνώ μαζί σου πάνω σε αυτό. Τώρα μερικά σχόλια σχετικά με τις τροπολογίες. Δεν ξέρω αν θα πρέπει ε, να δώσουμε χρόνο αγόρευσης ανάλογα με το μέγεθος ε, της έκθεσης, ε, αλλά δεν πειράζει. Σχετικά με την τροπολογία 1, παρόλο που τα κείμενα, τα ευρωπαϊκά μιλάνε πάρα πολύ για την Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Ένωση. Τι είναι, τι είναι. Είναι στην κάτι που είναι στη συνθήκη, διότι αυτό δεν είναι δημοσιονομική ένωση. Η φορολογική θα πρέπει να δούμε περί τίνος πρόκειται. Είναι νομίζω διφορούμενα τα πράγματα. Δεύτερον, τροπολογία 2 νομίζω αποδυναμώνει το κείμενο. Είναι για την ανταλλαγή πληροφοριών. Προτιμούμε το αρχικό κείμενο της Επιτροπής. Τροπολογία 5 ε, συμφωνώ με τον κύριο Κάζα εκεί όπου λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή. Εδώ μας λέει ο Νταβίδ, τα κράτη-μέλη καλούνται να ε, επικοινωνήσουν. Εμείς θα λέγαμε όχι are invited to, αλλά shall να είναι μια υποχρέωση. Θα βεβαίως θα υποβάλουμε γραπτό στις αλλαγές. Έχουμε ε, το κεφάλαιο 2 για το αίτημα ε, να μην υπάρχει μια γλώσσα ούτως ώστε να δοθεί έτσι μια πρόφαση στα κράτη-μέλη να μην πληρούν την υποχρέωση συνεργασίας. Δεν πρέπει να υπάρχουν παραθυράκια τα οποία θα ε, παρεμποδίζουν αυτή τη συνεργασία. Για το κεφάλαιο 3 ίσως θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τον κατάλογο των ε, αντικειμένων που θα μπορούσαν να περιληφθούν στις ανταλλαγές πληροφοριών. Αυτό που είπε όλε για την αρχή, την ευρωπαϊκή για τον ΦΠΑ, είπε ότι θα χρειαστούμε μια εισήγηση της Επιτροπής ε, για τις απάτες στον τομέα των εμέσων φόρων καταλώσεων. Ε, βεβαίως για το 2012 το θέλουμε αυτό. Είναι βραχυπρόθεσμο, είναι μικρή η προθεσμία, αλλά επειδή έχουμε διάφορα στρίπες στα δημόσια οικονομικά των κρατών θα πρέπει να δούμε τι φοροδιαφυγή υπάρχει γρήγορα διότι κάθε χρόνο είναι απώλεια εσόδων. Όσο πιο γρήγορα κινηθούμε τόσο καλύτερα θα μπορούμε ε, να έχουμε φορολογικά συστήματα πάνω σε υγιή βάση. Αυτά είναι προτάσεις και σχόλια και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Ashley. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που παρουσιάσατε κύριε Μίτσελ την έκθεση Κάζα. Είναι μια τεχνική έκθεση, δεν παρουσιάζει πολιτικά προβλήματα, είναι αποδεκτή ε, πολλής από την ε, ομάδα μου. Ενημερώνουμε κατά κάποιο τρόπο την έκθεση, την έκφραση και παίρνουμε περισσότερα στοιχεία μετά από την εισαγωγή του EMCS. Υποστηρίζουμε την έκθεση Κάζα, θεωρούμε ότι οι τροπολογίες του είναι λογικές ενισχύουμε και εμείς από πλευράς μας την πρόταση και θέλουμε πράγματι να προχωρήσει η διαδικασία την οποία στηρίζουμε πλήρως. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Υπάρχει ένα τεχνικό θέμα που απαιτεί διευκρινήσεις. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Γκέι, θες να ακούσουμε την Επιτροπή. Όχι, αν θέλουν κάτι βέβαια να πούν, Φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία για την έκθεση αυτή, μόνο αν υπάρχει κάτι το ζωτικό, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε το λόγο. Όχι να σχολιάσουμε, απλά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που θέσατε το θέμα σε συζήτηση τόσο γρήγορα. Είναι καλή η έκθεση, είναι θετικά τα σχόλια που ακολούθησαν και θα μεταφέρουμε φυσικά την έκθεση και τις προτάσεις σας προς την Προεδρία κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε. Γκέι, θες ξανά το λόγο. Σύντομα, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη για τη συμμετοχή του στην έκθεση Κάσα. Ο κύριος Κάσα θα είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την στήριξη. Θα μεταφέρω και τα σχόλια που έγιναν στον κύριο Κάσα. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει με το θέμα των αρχών για το ΦΠΑ. Όλα αυτά θα τα σημειώσω προς τον κύριο Κάσα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Πράγματι είναι πολύ τεχνική και μη προβληματική η έκθεση. Καλώ σας ευχαριστώ. Σας θυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία είναι η 1η Φεβρουαρίου. 12η Μεσημβρινή. Η εξέταση θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου και ελπίζω να φτάσουμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου υπαριθμών 2. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Πάξα. Ναι, ναι, α, δεν τον βλέπω, αλλά είναι στο βάθος. Πρόκειται για το σημείο 17, τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου. Για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δίνω τον λόγο στον εισηγητή. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι μάλλον σύντομος. Υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής που έρχεται σε μια στιγμή όπου ε, τα δημόσια οικονομικά είναι σε δύσκολη κατάσταση και οι δημόσιοι πόροι σπανίζουν. Έχουμε διάφορα έργα υποδομών, διάφορα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να προωθήσουν την οικονομία και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις τροπολογίες μου, τις οποίες ε, ε, συνέταξα αφού διαβουλεύτηκα διάφορους ενδιαφερόμενους. Έχουμε τα κράτη-μέλη τα οποία λόγω μεγάλων προβλημάτων χρηματοοικονομικής σταθερότητας έχουν ήδη λάβει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα μέσα επιμερισμού κινδύνων ε, να είναι διαθέσιμα για όλα τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν. Όχι μόνο για τα κράτη που έχουν δυσκολίες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, αλλά επίσης και οι χώρες ε, οι οποίοι έχουν ε, δυσκολίες ε, στην ιδιωτική χρηματοδότηση μεγάλων έργων δημόσιου ωφέλους που μπορεί να έχουν και δυσκολίες στο μέλλον. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να, το, να επιφέρουμε τροπολογίες συνεχώς του κανονισμού. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Η δεύτερη μου τροπολογία, η ιδέα πίσω από αυτή την τροπολογία είναι να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν, που χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά, να τα χρησιμοποιούν όχι μόνο ε, σε σχέση με τα έργα ε, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά και για άλλα μεγάλα έργα τα οποία προωθούν ε, την οικονομία και την απασχόληση. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για ε, σημαντικά έργα υποδομών ε, που ε, αποφέρουν εισόδημα, διότι τα άλλα δεν έχουν δυσκολία να προσελκύσουν ιδιωτική χρηματοδότηση. Αυτά που έχουν δυσκολίες πρέπει να βοηθηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αλλά η κατάσταση βλέπουμε ότι έχει αλλάξει σημαντικά και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να διευρύνουμε τον κανονισμό για να καλύψουμε επίσης αυτά τα έργα. Αυτό το μέτρο είναι προσωρινό, θα ισχύει μόνο μέχρι το τέλος του, του, της προγραμματικής περίοδου. Ήδη τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν τη νέα προγραμματική περίοδο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερνικήσει την κρίση και νομίζω ότι η Επιτροπή αφού αξιολογεί στην επιτυχία αυτών των μέτρων θα μπορούσε να προτείνει μόνιμα μέτρα. Ελπίζω να βρείτε αποδεκτές τις τροπολογίες μου και περιμένω να ακούσω τη γνώμη σας και τις προτάσεις που θα διευκολύνουν την υλοποίηση και εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ σύντομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την Qui Και στην Επιτροπή ΙΤΡΕ και είναι εισηγητή για το θέμα που συζητείτε τώρα. Θα κοινοποιήσω στον εισηγητή τις παρατηρήσεις του κυρίου Καρίνς που είναι πάρα πολύ τεχνικές επειδή δεν γνωρίζω το φάκελο αυτό. Φοβούμαι μήπως πω ανοησίες Γι' αυτό θα δώσω τις σημειώσεις αυτές στον εισηγητή που θα τις ε, χρησιμοποιήσει με κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του αλλά νομίζω ότι εφόσον η Επιτροπή είναι παρούσα, θα επωφεληθώ για να θέσω ερωτήσεις στην Επιτροπή. Πρωτού προχωρήσουμε σε αυτήν την εργασία, θα ήθελα διευκρινήσεις για ορισμένα σημεία. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τα έργα αυτά. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση, διότι από ό,τι κατάλαβα, νομίζω ότι κατάλαβα, το χρονοδιάγραμμα στην Επιτροπή Ρέτζι είναι έχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ισχύει αυτό, είναι αλήθεια. Και θα ήθελα να μάθω εάν η πρόταση του εισηγητή και η πρόταση διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής αυτού του κειμένου, όχι μόνο για τις χώρες που αποτελούν μέρος του προγράμματος, αλλά και στους άλλους, όχι μόνο στα ταμεία συνοχής, αλλά και στα άλλα ταμεία, τι επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι προτάσεις σε σχέση με την αντίληψη που είχε αρχικά η Επιτροπή. Και θα ήθελα επίσης να μου πείτε εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη διεύρυνση της διαδικασίας που προβλέπεται για την Ελλάδα για να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες του προγράμματος λόγω της κατεπίγουσας κατάστασης, γιατί μου φαίνεται ότι ο μηχανισμός αυτός είναι ενδιαφέρον μηχανισμός και ότι στην εκπόνηση της θέσης μας θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι, ποιοι είναι οι όροι βιωσιμότητας που θα προταθούν. Επιφυλάσσω λοιπόν τη θέση μου, ενώ δεν θα έχω καταλάβει καλύτερα τη θέση της Επιτροπής σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, σχετικά με τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής για άλλες χώρες, ε, του προγράμματος και για το σύνολο των χωρών. Εάν η πρόταση λοιπόν του συναδέλφου μου είναι βιώσιμη η πρόταση στα μάτια της Επιτροπής. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να έχω αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ κυρία Φερέρα. Uh, αυτό το θέμα του επιμερισμού κινδύνου ε, με εξέπληξε αυτό και διαρωτώ με πού σταματάει ο κίνδυνος και που έχουμε μια πραγματική αξιολόγηση του κίνδυνου. Όλοι Σμιτ στην ε, ε, προηγούμενη εισήγηση είχε πολύ λίγο χρόνο πριν τη συζήτηση. Εγώ α, ε, είχα περισσότερο χρόνο. Χθε το απόγευμα ορίστηκα σκιώδη συγκητή. Έτσι γίνονται τα πράγματα σε ορισμένε ομάδε. Έχω κάποιο σκεπτικισμό σχετικά με τη σημερινή συζήτηση ίσως είναι ανταμοιβή για τις χώρες που διαχειρίζονται άσχημα τις οικονομίες τους. Θα επανέλθω ίσως αργότερα με πιο ενδελεχή στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καμάλ. Ο σκιώδης εισηγητής τώρα της ΑΛΤΕ, ο κύριος Κυλακάκης παρακαλώ. Συγγνώμη για την κακή προφορά του ονοματός σας. Έχετε τον λόγο κύριε Σκυλακάκη ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα η οικονομική κατάσταση γενικά στις χώρες στις οποίες αναφερόμαστε είναι τελείως διαφορετική από τότε όταν σχεδιάζαμε το στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για αυτές. Έχουμε ένα νέο κόσμο μπροστά μας στην Ελλάδα για παράδειγμα και σε κάποιο βαθμό και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία και πρέπει να μεταθέσουμε κονδύλια, χρήματα σε αυτόν τον νέο κόσμο να ε, υπάρξουν αυτές οι δράσεις. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό σε αυτόν τον νέο καινούριο κόσμο. Κανείς τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν αναλαμβάνει νέα οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι πολίτες δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι το νόμισμα αύριο και έτσι δεν κάνουν επενδύσεις ούτε καν λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Και αυτό θα διαρκέσει κατά τον ένα ή άλλο τρόπο με, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας τρόπος να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις. Και αυτό είναι μια πολύ καλή οδός να κάνουμε, να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Εμείς στην ομάδα της Άλντε προτείναμε μια παρόμοια ε, δράση όπως αυτού του μέσου τον Ιούνιο ήδη του 2011 και με ικανοποίηση βλέπουμε ότι έλαβε υπόψη και μάλιστα με θαραλέο τρόπο και θαραλέο διάβημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό Τώρα, αν αυτό θα είναι χρήσιμο μέσο για άλλε χώρε ή όχι, είμαστε ανοιχτοί και πρέπει να το δούμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμω ότι το χρονοδιάγραμμα, timetable, έχει τεράστια σημασία. Πρέπει να υλοποιηθεί το δυνατόν γοργότερα αυτό το χρονοδιάγραμμα. Επειδή θα βοηθήσει το σύνολο τη Ευρώπη, αν σταθεροποιηθούν αυτέ οι χώρε με τι δράσει μα. Και οι επενδύσει, ιδιαίτερα επενδύσει του ιδιωτικού τομέα, που θα έχουν μία, έναν ε, κοινό ε, κίνδυνο που θα συμμερίζονται όσοι θα εμπλέκονται, είναι κάτι που μπορεί να συμπράξει στην σταθεροποίηση των αγορών. Χρειάζονται τέτοια θετικά μηνύματα που πρέπει να αποστείλουμε. Τώρα, δύο πράγματα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε μέσα στο πλαίσιο αυτού του νέου κανονισμού. Το ένα είναι ότι αυτά τα χρήματα θα περάσουν σε ένα απόλυτα νέο καινοτόμο μέσο το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα. Θα είναι άδικο λοιπόν και αθέμητο να απολεστούν αυτά τα κονδύλια αν χρειαστεί κιόλα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την κινητοποίηση αυτού του μέσου. Ιδιαίτερα όταν γίνεται στο παραπέντε, το τελευταίο λεπτό στο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, ελαστικοί για το πώ θα γίνουν αυτά. Πώ δηλαδή τα χρήματα θα διατεθούν και θα τα διαχειριστούμε μετά το τέλος δηλαδή ε, την εκπνοή αυτού του μέσου, αυτού, αυτής της διευκόλυνσης. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι πρέπει να συντάξουμε, να καταρτήσουμε ένα κανονισμό που θα μπορεί να γεφυροποιήσει τα δύο αυτά πλαίσια. Δεν έχουμε πλέον άλλο χρόνο για να συντάξουμε, να καταρτήσουμε ένα νέο κανονισμό ή να αλλάξουμε και να προσαρμόσουμε τον κανονισμό περνώντας στη νέα δημοσιονομική περίοδο. Αυτό το πράγμα θα αρχίσει να λειτουργεί, θα είναι λειτουργικό μετά από 6 μήνες ας πούμε από σήμερα και πρέπει να διαρκέσει για παραπάνω από ένα έτος ή ενάμιση έτος. Εντάξει, τούτων λεχθέντων πρέπει λοιπόν, χρειάζεται να έχει ένα μεγαλύτερο διάστημα εφαρμογής και να είναι ασφαλέστερο για τις χώρες που θα εμπλέκονται. Το να πάρουμε χρήματα από δημόσια τέτοια προγράμματα και σχέδια που θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί σήμερα και να τα εντάξουμε στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων κατά το μεγαλύτερο βαθμό ή για περισσότερα δημόσια τέτοια προγράμματα Μειώνοντα τον κίνδυνο, αυτό είναι ακριβώ αυτό που κάνουμε, μειώνουμε τον κίνδυνο, πρέπει να είμαστε ελαστικοί, ευέλικτοι σε αυτό. Ευχαριστώ. Uh, Σα ευχαριστώ πολύ. Ο Φιλίπ παρακαλώ. uh... Συμφωνώ με το ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη σήμερα κοινοτοποίηση της ιδιωτικής επένδυσης σήμερα. Οι επενδυτικές δυνατότητες στην Ευρώπη βρίσκονται στα χέρια των οικοκυριών και μη ε, πιστοτικών ιδρυμάτων. Αυτό το χρήμα πρέπει να το κινητοποιήσουμε. Να κινητοποιήσουμε λοιπόν τις επενδύσεις αυτές είναι κάτι το αυτονόητο. Έχουμε δύο όμως ε, προϋποθέσεις που συνδέονται με την ιστορία των διαφορετικών ταμείων. Το πρώτο είναι γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά. Είδαμε στην Πορτογαλία και αλλού Νομίζω ότι ο τρεμός από τους φιλελεύθερους είχε αναφερθεί στον αριθμό των αεροδρομίων που χτίζονται στην Ισπανία και όπου δεν απογειώνεται κανένα αεροπλάνο από τα αεροδρόμια αυτά. Και γνωρίζουμε πόσο οι υποδομές αυτές δεν ήσαν οικονομικά υποστηρίξιμες, αλλά χρηματοδοτήθηκαν με τα διαφορετικά ταμεία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει εδώ μια ανάγκη για αλλαγή πορείας σε σχέση με αυτά. Να περιμένετε λοιπόν τροπολογίες από πλευράς μας, οι οποίες θα στηρίξουν την αιρεσιμότητα, την αρχή της αιρεσιμότητας και τον έλεγχο του τι έγινε με τα χρήματα αυτά, ακόμα και αν λειτουργούν σαν καταλήτες για ιδιωτικές επενδύσεις και κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Στην Πολωνία, σαν παράδειγμα, κάποια προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση ήταν παράνομα σε σχέση με τον κανονισμό Natura 2000. Αυτό δεν μπορούμε να το στηρίξουμε πλέον. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω όλες αυτές οι επενδύσεις να μοχλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καταστήσουν τις οικονομίες πιο αηφόρες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, σαν παράδειγμα, ε, η παραβίαση των κανόνων για το περιβάλλον μειώνει την ε, έλξη την οποία ασκεί σαν τουριστική χώρα ε, η Ελλάδα. Τώρα, η διαφάνεια των διαδικασιών. Νομίζω ότι η εμπλοκή γύρω από τις επιλογές μάλλον ή ε, ε, τις πολιτικές γύρω από αυτά τα προγράμματα μένουν πολλά να γίνουν. Το Κοινοβούλιο σχετικό με το πολιετές πλαίσιο έχει θα έλεγα κάνει κάποιες προτάσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τις δυνατότητες επιλογής των προγραμμάτων. Έχει ζητήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η EID τον λόγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει, θα έλεγα εδώ, προτεραιότητα. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει πρώτος. Η Επιτροπή μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πολύ συγκεκριμένο μέσο για μια πάρα πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Το μέτρο αυτό αντιμετωπίζει τα σημαντικά εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες και σε αυτή τη φάση η Ελλάδα για την έβρεση ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων έτσι ώστε να προωθηθούν κάποια προγράμματα υποδομών που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο χρήμα μόνο εν μέρη. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία θα προσφέρουν κέρδος σε μια χρονική περίοδο και που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως από δανειοδοτήσεις μέσω των Ταμείων Συνοχής. Το μέγιστο ποσοστό ε, θα έλεγα ελέγχεται ε, συμμετοχής της κοινοτικής βοήθειας ε, συμπληρώνεται και από τους κανόνες τους εθνικούς. Είναι απαραίτητο λοιπόν να συνδεθεί το τμήμα του προγράμματος το οποίο χρηματοδοτείται κανονικά από τον δημόσιο τομέα με τα μέσα τα κοινοτικά, από τα κοινοτικά ταμεία και με το κομμάτι το οποίο χρηματοδοτείται απευθείας από τους ιδιώτες <clears throat> και θα αποσβέσουν οι ιδιώτες μέσω των μελλοντικών κερδών που θα σημειώσουν οι υποδομές. Σήμερα όμως δυστυχώς στην Ελλάδα, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και σε άλλες χώρες, οι οποίες επηρεάζονται από την κρίση, οι ιδιώτες επενδυτές δεν έρχονται μπροστά, δεν διακινδυνεύουν και δεν ξεκινούν δυστυχώς τα συγκεκριμένα προγράμματα. Κάποια από τα στρατηγικά αυτά προγράμματα, τα οποία έχουν επιλογή, είναι σε κίνδυνο και κινδυνεύουν ακριβώς να μην εφαρμοστούν γιατί δυστυχώς ε, ο ιδιωτικός τομέας είτε δεν έχει αυτή τη στιγμή τη ρευστότητα, είτε δεν έχει τη διάθεση να επενδύσει στα πλαίσια των σημερινών συνθήκων. Το μέτρο το οποίο προτείνεται λοιπόν είναι πραγματικά ένα μέτρο κατανομής αν θέλετε κινδύνων γιατί μεταφέρει κατά κάποιο τρόπο προς τα κράτη-μέλη πόρους οι οποίοι συχματοδοτούνται από τα διαφορετικά ταμεία και μεταφέρει και ένα τμήμα του κινδύνου τον οποίο κανονικές αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας υπό ΚΣ, σήμερα όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας δεν το κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Πώς μπορεί τώρα το μέτρο αυτό να εφαρμοστεί. Μπορεί να εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτημα του συγκεκριμένου κράτους μέλους σε συνεργασία με το EIB ή με κάποια άλλο εθνικό ή διεθνές σώμα το οποίο έχει σαν αποστολή να παρέχει εγγυήσεις όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα έχει θα έλεγα μια παράδοση στον τομέα αυτό συμμετοχή στην ανάληψη ευθυνών σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να χρηματοδοτούνται προγράμματα συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία και με τους στόχους της κοινοτικής πολιτικής. Το συγκεκριμένο κράτος μέλος λοιπόν θα πρέπει να καταθέσει μια επίσημη αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει τα προγράμματα και τις επενδυτικές ανάγκες τις οποίες θα ήθελε να καλύψει στα πλαίσια ακριβώς του μέσου κατανομής κινδύνων τέτοιου είδους χρηματο, ε, χρηματοδοτικές ανάγκες δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερες από τη διαφορά ανάμεσα στο προβλεπόμενο κόστος και στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό ε, χρηματοδότησης από πλευράς των ε, Ταμείων Συνοχής. Έχουμε ξεκάθαρη πρόθεση τα μέσα αυτά να μην χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν το χρέος της συγκεκριμένης χώρας, αλλά να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να επιτρέπουν κάποια προγράμματα τα οποία ήδη συγχρηματοδοτούνται από τα διαθροτικά ταμεία να χρηματοδοτούνται μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό συγχρηματοδότησης σύμφωνα με τον κανονισμό των ταμείων και με τον κανονισμό των, των, των αντίστοιχων που ισχύει στη συγκεκριμένη χώρα. Γιατί οι εθνικές ρυθμίσεις μερικές φορές προβλέπουν να μην ξεπερνούμε κάποια επίπεδα. Λοιπόν, στόχος του μέτρου είναι να γεφυρωθεί το κενό αυτό το οποίο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί σήμερα γιατί δεν προσέρχεται θα έλεγα να καλύψει την ανάγκη ο ιδιωτικός τομέας. Το κράτος μέλος λοιπόν θα πρέπει να εντοπίσει τα προγράμματα, θα πρέπει να δει τους πόρους τους οποίους μπορεί να διαθέσει στο μέσο αυτό κατανομής κινδύνων. Το κράτος θα πρέπει να εντοπίσει σωστά ποιες είναι οι ανάγκες και ποιοι είναι οι πόροι οι οποίοι θα περάσουν από τα υπάρχοντα προγράμματα στο συγκεκριμένο αυτό μέσο και να αξιολογήσει την ανάγκη η οποία υπάρχει έτσι ώστε να προχωρήσουν τα προγράμματα αυτά. Από την άλλη, το κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλει το πρόγραμμα στο, ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή σε κάποιο άλλο χρηματοπιστωτικό όργανο το οποίο μπορεί να παίξει τον ίδιο ρόλο και έχει την ίδια αποστολή έτσι ώστε να υπάρξει συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λοιπόν θα πρέπει να κάνει τη λεγόμενη due diligence σε σχέση με το πρόγραμμα να εξετάσει οικονομικά και χρηματοδοτικά την βιωσιμότητα του προγράμματος, έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμο ακριβώς το πρόγραμμα αυτά και να μην χρηματοδοτηθούν μη βιώσιμα προγράμματα. Γιατί δίδονται δάνεια από πλευράς ε, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν, θα πρέπει να αποσβεθούν. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο γιατί έχουμε μία ακρόαση η οποία ακολουθεί τώρα. Δευτερόλεπτα και κλείνω. Επί τη βάση λοιπόν του αιτήματο από πλευρά του κράτου μέλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει μία απόφαση εγκρίνοντας τη μεταφορά πόρων από τα υπάρχοντα προγράμματα στο συγκεκριμένο μέσο. Και μια τέτοια απόφαση θα ορίζει και τις συνθήκες κατά από τι οποίες το συγκεκριμένο μέσο θα τεθεί σε λειτουργία. Παραδείγματα σήμερα Έχουμε την δανειοδοτική ε, και εγγυητική διαδικασία ή μέσο αν θέλετε για την περιοχή του Δούναβη. Έχουμε επίσης ε, και την αντίστοιχη διαδικασία που προβλέπεται για το 7ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο. Βλέπουμε εδώ πως μοιραζόμαστε τον κίνδυνο με τον ιδιωτικό τομέα και εμπνεόμεθα από αυτό σε σχέση με τον χρονισμό όπως ε, το ζήτησε το συγκεκριμένο μέλος. Κοιτάξτε. Εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε. Και τώρα ε, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα ήθελε να παρέμβει. Πολύ σύντομα, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, σίγουροι είμαι ότι... Κοιτάξτε, δεν θέλω κατηδίαν συζητήσεις, Φιλίπ, εντάξει, στην αίθουσα. Λοιπόν, ο χρόνος έχει πλέον λήξει. Ποιος θα παρέμβει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πραγματικά δεν έχουμε πλέον χρόνο για ε, μακρηγορίες από πλευράς της, ε, ε, των ομιλητών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα είμαι πολύ σύντομη η ΕΤΕΠ καλωσορίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύει ότι η δημιουργία αυτού του ειδικού μέσου θα μας επιτρέψει να παράσχουμε χρηματοδότηση για έναν αρκετά μεγάλο αριθμό προγραμμάτων και σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σε μια χρονική συγκυρία όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου η ρευστότητα του χρηματοοικονομικού τομέα σπανίζει και ζητήθηκε η αύξηση συμμετοχής για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμματών υποδομών. Αυτό το μέσο συμμετοχής στους κινδύνους θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην απορρόφηση των διαθωτικών κονδυλίων τώρα που προσεγγίζουμε την ολοκλήρωση. Και επίσης υποστηρίζουμε το σχέδιο έκθεσης που προετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια και έχουμε και δύο προτάσεις εδώ που ε, την χάνουν διαφοροποίησης, πρέπει να τύχουν διαφοροποίησης σε σχέση με την ε, μη χρηματοδότηση δράσεων από την ΤΕΠ και το ε, Ταμείο Συνοχής που όμως έχουν μεγάλη σημασία για το κράτος μέλος και πρέπει να δίνεται η εναλλακτική λύση στα ίδια τα κράτη-μέλη αν θέλουν να λειτουργήσει αυτό το μέσο με αυτόν τον τρόπο ή όχι. Θα επιτρέψει λοιπόν αυτό το μέσο για τα διαθροτικά ταμεία να έχουν μια μεγαλύτερη επίπτωση, θετικότερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ πολύ, λέγει Πρόεδρος. Η κυρία Κλέβερ είχε ζητήσει να παρέμβει. Απλά να αποσαφηνίσω ήθελα σε σχέση με την Επιτροπή Περιφερειακών Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ναι, έχουμε όμως μια ακρόαση στην οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Πολύ σύντομα επανερχόμεθα στον εισηγητή αν θέλει να κάνει κάποια σχόλια για όλα τα άλλα θέματα, αν η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλει να αναφέρει κάτι στα μέλη, μπορούν γραπτώς να το διαβιβάσουν στη γραμματεία μας και η γραμματεία θα διασφαλίσει ότι θα διανεμηθούν ε, αυτές οι παρατηρήσεις και σημειώσεις ε, στους ε, εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές. Εσείς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Όλα τα μέλη που συνεισέφεραν και εξέφρασαν τις απόψεις τους τα ευχαριστώ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΕΛΚΑ που υποστήριξαν την πρότασή μου και ευχαριστώ και εκείνους που ήταν λιγότερο αισιόδοξοι, ας το αποκαλέσω έτσι, σε σχέση με την έκθεση αυτή. Όλες οι προτάσεις σας θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων ούτως ή άλλως. Δύο πράγματα θέλω να πω. Ε, ε, σε σχέση με την συσσόρευση επαρκούς πείρας για τη διαχείριση παρόμοιων προγραμμάτων όσον αφορά ε, τη διαχείριση ζητημάτων για την έρευνα και ανάπτυξη, ένα άλλο θέμα το οποίο πιστεύω ότι όλα τα μέλη πρέπει να υποστηρίξουν σε αυτή τη συνεδρίαση είναι το ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την προαγωγή των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η κύρια προτεραιότητά μας, ούτως ή άλλως. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που είναι διαθέσιμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης θα είναι 24 Ιανουαρίου, δηλαδή σήμερα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η 10η Φεβρουαρίου. Εξέταση και έγκριση με ψήφιση ε, των τροπολογιών. Ε, Πολλέ ε, είναι οι ημερομηνίε εδώ, έτσι. Λοιπόν. Α, μάλιστα. εντάξει, αυτό εξαρτάται από τι θα συμβεί στην επί τη ουσία αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ω ημερομηνία. Θα πρέπει να αναμείνουμε λοιπόν από σαφήνιση αυτή τη ημερομηνία στη συνέχεια εν ευθέτω χρόνο. Και περνάμε τώρα στη συνέχεια αμέσω στο θέμα της κρατικής, του κρατικού χρέους. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση Προέδρου. Ίσως κάποιοι γνωρίζετε, αναμένουμε την τελική απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων για την σύνταξη έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας που ζητήσαμε να συντάξουμε για την προσπελασιμότητα στο Basic Banking. Ζητήθηκε και από την Ίνκο να συνταχθεί μια τέτοια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας θα συνέλθουμε για να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό πριν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το θέρος. Έχουμε καθορίσει ένα προσωρινό σχεδιάγραμμα εξαρτώμαστε από την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων ποια θα είναι επί της ουσίας αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και φαίνεται ότι θα είναι στις αρμοδιότητες της ΕΚΟΝ όπως έχουν τα πράγματα. Παρουσίαση της σχεδίου έκθεσης 12 Μαρτίου στο Στρασβούργο προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 22 Μαρτίου και έκθεση και ψήφιση τροπολογιών 24 και 25 Απριλίου με στόχο να ψηφίσουμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Επιτροπή 30-31 Μαΐου να καταλήξουμε στην περίοδο συνόδου στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Αυτό είναι το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για όσους ενδιαφέρονται γι' αυτό. Πολλές συζητήσεις διεξάγονται στην αίθουσα. Όσοι θέλουν να συζητήσουν αναμεταξύ τους να αποχωρήσουν εκτός αίθουσας. Παρακαλώ. Because we now wish to... τώρα θα, θέλουμε, θα θέλαμε να προχωρήσουμε στη δημόσια ακρόαση, αν γίνεται. Okay. Right. Okay. Um, this is the second part. Είναι το δεύτερο τμήμα αυτό της ε, ακρόασης που είχαμε κατά το, ε, τη χθεσινή ε, ημέρα. Είχαμε κάποιους ε, πραγματογνώμονες εχθές παρόντες. Υπήρξε και η απουσία τους λόγω της διεξαγωγής της συνάντησης του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ και δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες εχθές όπως είχε προβλεφθεί και είναι σήμερα παρόντες. Γι' αυτό έχουμε σε δύο σκέλη αυτή την ακρόαση. Σκοπός της ακρόασης είναι, σας υπενθυμίζω, να εξετάσουμε... Συγγνώμη, δεν μπορώ να συναγωνιστώ με τις κατηδίαν συζητήσεις των μελών ο στόχος και το νόημα αυτής της ακρόασης είναι και ήταν διακόπτη πρόεδρος. Δεν μπορώ να ανταγωνιστώ με τις άλλες συζητήσεις. Ελίζα, παρακαλώ, σταματήστε τις συζητήσεις. Αν θέλετε να παραμείνετε, επειδή δεν θα είναι δυνατόν να συνεχίσουμε και να παραμείνετε περισσότερο στην αίθουσα, εντάξει τότε. Λοιπόν, σταματήστε αν γίνεται. Ευχαριστώ. Στόχος και σκοπός αυτής τη ακρόασης είναι να εξετάσουμε τα τρέχοντα ε, σε ισχύ μέσα και εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρατικής υπερχρέωσης όπως τη Ελλάδα και την αντιμετώπιση των μέσων που έχουν σχεδιαστεί και των επιπτώσεων για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα με τη χρήση του μέσου ε, οικονομική νομισματική σταθεροποίηση. Επίσης ε, για τη χρήση του ESM, πότε θα αρχίσει να λειτουργεί και όλα τα συναφή αυτά θέματα. Με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να πω ότι έχουμε ανάμεσά μας τον Klaus Regling, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESFS. Ε, και επίσης ε, έχουμε και τη Γενικό Διευθυντή ανάμεσά μας του ECOFIN. Με όλους αυτούς λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ρέγκλινγκ. Σωστό Μάλιστα. Ίσως μπορείτε να μας ενημερώσετε λοιπόν για την κατάσταση σε σχέση με το πώς έχουν τα πράγματα και όπως τα βλέπετε θα περάσουμε μετά στον κύριο Γκούτι και, μετά... Μπούτι και θα έχουμε τη συζήτηση με τα μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας μιλήσω για το δικαίωμα μου τομέα ε, αρμοδιότητας, ε, το EFSF και την προετοιμασία του EFSM και ο Μάρκο Μπούτι θα σας ε, μιλήσει για το EFSM ε, και τα άλλα θέματα σε σχέση με τον προϋπολογισμό, τον κοινοτικό και τις επιπτώσεις της χώρας, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσα στις χώρες. Τι έχει κάνει το EFSF μέχρι τώρα από τότε που δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2010. Υποστηρίζουμε δύο προγράμματα προσαρμογής Αυτά τα δύο προγράμματα υποστηρίζονται από το EFSF, EFSM, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και διάφορες συνεισφορές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Ε, το EFSF υποστηρίζει τα τρία Ιρλανδικά προγράμματα με 17,7 δισεκατομμύρια και τρία προγράμματα πορτογαλικά με 26 δισεκατομμύρια για να το κάνει αυτό μέχρι τώρα έχουμε εκδώσει ομόλογα μακροπρόθεσμα με ορίμανση 3, 5, 10 ετών που καλύπτουν 22 δισεκατομμύρια. Δεν είχαμε καθόλου προβλήματα για τα ομόλογα αυτά στην αγορά και πριν από δύο μήνες εκδώσαμε μερικά γραμμάτια, 11 γραμμάτια. Και και 9 ε, εκατομμύρια στην Πορτογαλία. Για το υπόλοιπο του έτους αυτό, 2012, θα εκταμιεύσουμε ακόμα 5 εκατομμύρια στην Ιρλανδία και 11 στην Πορτογαλία. Βεβαίω αυτό πάντοτε υπό την αίρεση της ανασκόπησης που θα κάνει η Τρόικα, δηλαδή η Επιτροπή, το Δούνου του και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτω ώστε οι προποθέσει να τηρηθούν, να έχουν ληφθεί τα μέτρα αναδιάρθρωση τη οικονομία που έχουν αναλυφθεί. Όταν άρχισε τον Μάιο-Ιούνιο 2010 το EFSF είχε ε, δυναμικότητα 240 δισεκατομμύριων ευρώ. Από τότε έχουμε προχωρήσει. Έχουμε ε, τώρα το EFSF 2 ε, με δυναμικότητα 440 δισεκατομμυρίων και νέα μέσα. Ε, γνωρίζετε ποια είναι αυτά τα νέα μέσα. Πρόκειται για παρεμβάσεις, αγορές στον πρωτογενή και δευτερογενή ε, τομέα ομολόγων, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών σε χώρες ε, που δεν έχουν ένα πρόγραμμα προσαρμογής γενικό. Όταν τα μέσα αυτά λειτουργούν καλά, τα κατευθυντήριε ε, γραμμές συμφωνήθηκαν τον Νοέμβριο, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα, διότι καμία χώρα δεν ζήτησε την χρήση των μέσων αυτών αλλά όλες οι τεχνικές προπαρασκευές και υποδομή υπάρχουν ήδη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας βοηθάει για την εφαρμογή κυρίως της αγορές στη δευτερογενή αγορά, αν απαιτηθούν και αν ζητηθούν. Επίσης, να σας μιλήσω για την μόχλευση των πόρων μας, διότι αυτό συζητήθηκε πολύ τους τελευταίους μήνες. Ίσως γνωρίζετε ότι έχουμε αναπτύξει ε, δύο επιλογές μόχλευσης όπου το EFSF εγγυάται ε, ανάμεσα σε 20-30% σε περίπτωση χρεοκοπίας. Η πρώτη ε, επιλογή είναι ένας τύπος ασφάλισης που έχει προετοιμαστεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν το ζητηθεί από μια χώρα. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα, τα τεχνικά, τα νομικά. Η δεύτερη επιλογή που είναι ένα ταμείο συνεπένδυσης ε, για χρήματα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι έτοιμο το μέσο αυτό και σε μερικές εβδομάδες θα μπορούσε να λειτουργήσει και θα απαιτούσε βεβαίως αίτηση από μια χώρα για να χρησιμοποιηθεί. Οι επενδυτές έχουν ανταποκριθεί αρκετά θετικά σε αυτές τις δύο επιλογές και είμαι πεπισμένος ότι και οι δύο αυτές επιλογές θα χρησιμοποιηθούν στην αγορά. Σχετικά με την δεύτερη επιλογή συνεπένδυσης έχουμε δεσμεύσεις από επενδυτές εκτός Ευρώπης που ανέρχονται σε 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως η δοκιμή, πώς θα πρέπει να δοκιμάσουμε πώς θα λειτουργήσουν στην αγορά τα μέσα αυτά και ε, πόσα ε, κεφάλαια μπορούν ε, να κινητοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν από αυτά τα μέσα μόχλευσης. Θα το δούμε αυτό όταν υπάρχει έτοιμα από μια χώρα. Διότι αν δεν υπάρξει έτοιμα και δεν χρησιμοποιηθούν, πώς θα δοκιμαστούν. Σχετικά με το EFSM, τον μόνιμο μηχανισμό που θα αρχίσει να λειτουργεί από τον Ιούλιο του επομένου έτους, το EFSF ανέλαβε να προετοιμάσει ε, το EFSM πριν από δέκα μήνες. Του ανατέθηκε το έργο αυτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και έχει τα μέσα, τα χρηματικά για να το πράξει, τους πόρους. Έχουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία, προσλαμβάνουμε προσωπικό, έχουμε όλα τα τεχνικά μέσα τα οποία απαιτούνται, συστήματα μηχανογράφησης, επικοινωνίας, πληροφορίας, όλα θα είναι έτοιμα τον Ιούλιο 2012, ένα χρόνο πριν από ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά, όπως αποφασίστηκε από την σύνοδο της 9ης Δεκεμβρίου πέρσι το Eurogroup και οι Υπουργοί Οικονομικών πέρσι οριστικοποίησαν τη συνθήκη για το EFSM που θα υποβληθεί στα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι σημαντικό επίσης να επισημάνω ότι η κεφαλαϊκή επάρκεια θα επανεξεταστεί τον Μάρτιο και αυτό είναι μια απόφαση που λήφθηκε από τη Σύνοδο Κορυφή το Δεκέμβριο. Αυτό είχα να πω και τώρα δίνω τον λόγο στον συνάδελφο Μάρκο Μπούτη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Επιτροπή ήταν πάρα πολύ δραστήρια στο να βοηθήσει για την προετοιμασία αυτών των αντιπυρικών μέσων και ζωνών. Έχουμε προσωπικό για το EFSF και εμείς συμμετείχαμε επίσης, εμπλακήκαμε στην παροχή τεχνικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό του μηχανισμού του μονίμου. Ε, ασχοληθήκαμε άμεσα με τρεις βασικούς ε, τύπους στήριξης. Πρώτο, η Ευρωπαϊκή Δανειακή Διευκόλυνση στην Ελλάδα, μετά η FSM και μιλάμε, δεν μιλάμε τόσο πολύ τελικά για το τρίτο πράγμα, αλλά είναι κάτι σημαντικό μια φάση της κρίσης που μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε ε, προβλήματα εκτός της Ευρωζώνης, δηλαδή προβλήματα ελλείμματος, προβλήματα αύξησης των μέσων για την, το ισοζύγιο πληρωμών. Περάσαμε στα 50 δισεκατομμύρια και το μέσο αυτό μας επέτρεψε παρέμβαση ε, στην Λετωνία, Ρουμανία, Ουγγαρία και έχουμε ακόμα 37 ε, ε, δισεκατομμύρια υπόλοιπο. Σχετικά με το δανειακό μέσο για την Ελλάδα, πρόκειται για δάνεια που παρέχονται διμερώς από τα κράτη-μέλη στην Ελλάδα. Τι κάνει εδώ η Κομισιόν έχει βασικά έναν καθαρό συντονιστικό ρόλο, δηλαδή ε, εγγυάται, εξασφαλίζει ότι τα χρήματα παρέχονται στον κατάλληλο χρόνο ε, και ε, ασχολείται με το επιτόκιο να μην είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο. Πρόκειται λοιπόν για τεχνική βοήθεια που παρέχουμε εδώ. Έχουμε πλήρη συμμετοχή και ευθύνη για την διαχείριση του EFSM. Θυμάστε ότι όταν δημιουργήθηκε το EFSF, αρχικά ήταν, δημιουργήθηκε επίσης με 60 δισεκατομμύρια με τον αρχική αντιπυρική δύναμη. Τώρα το EFSM έχει 48,5 δισεκατομμύρια δεσμευμένα, υπάρχουν, έχει εκταμιεύσει 31 και η Επιτροπή εκ, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει επίσης ε, περάσει σε έκδοση ομολόγων από ε, κεφάλαια που έχουν παρασχεθεί και που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα 27 κράτη-μέλη. Όπως ε, επεσήμενε η κυρία Πρόεδρος, το μηχανισμό CFSM έχει υποστήριξη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το θέμα που τίθεται είναι ένα από τα ερωτήματα που θέσατε στην ημερήσια διάταξή σας. Ε, ε ποια θα είναι επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό τον κοινοτικό όταν χρησιμοποιηθεί ο EFSM. Όλα τα δάνεια στους δικαιούχους ε, χρηματοδοτούνται σε, με βάση back-to-back, -back, to back δηλαδη με ομόλογα και δεν αναλαμβάνεται κανένα κίνδυνο όσο προ τη διάρκεια και προ το επιτόκιο. Δανειζόμαστε χρήματα στην αγορά και μετά τα κεφάλαια αυτά πηγαίνουν στου δικαιούχου. Ο μόνο κίνδυνο που έχουμε είναι ένα credit risk, δηλαδή εάν βεβαίω ο δικαιούχο δεν εξυπηρετήσει το δάνειο αυτό, δεν τηρήσει τι υποχρεώσει των τοκοχρεωλησίων. Υπάρχουν ορισμένες βαλβίδες ασφαλείας για να εξασφαλίσουμε ε, να μην ε, πραγματοποιηθεί ο κίνδυνος, να μην υλοποιηθεί πρώτα απ' όλα. Υπάρχουν ε, δάνεια τα οποία οφείλονται 14 ημέρες πριν από την ορίμανση του ομολόγου. Δηλαδή αυτές οι 14 μέρες είναι μια βαλβίδα ασφαλείας για παρέμβαση σε περίπτωση που υπάρχει αθέτηση πληρωμής, εάν δεν έχει αποπληρωθεί όπως έπρεπε το δάνειο. Βεβαίως δεν περιμένουμε να συμβεί μια τέτοια περίπτωση. Εάν αυτή, αυτό το, το, η βαλβίδα ασφαλείας δεν αποφέρει καρπούς. Υπάρχουν και άλλες βαλβίδες που υπάρχουν στο νομικό, δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτως ώστε η, η Επιτροπή να μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές. Ο Κλάους ε, ε, ανέφερε πού βρισκόμαστε στο EFSF, στο EFSM εμείς ε, χρησιμοποιούμε τους σπόρους αυτούς σε συνδυασμό με το EFSM για χώρες του προγράμματος ε, για την Ευρωζώνη. Πού βρισκόμαστε σχετικά με τα προγράμματα αυτά. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Ελλάδα. Ανέφερα ότι η βοήθεια στην Ελλάδα ε, για την Δανειακή Σύμβαση του Μαΐου 2010 είναι 110 δισεκατομμύρια 80 από την Ευρωζώνη και 30 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διαβάζετε τον τύπο, παρακολουθείτε το θέμα. Τώρα ε, διαπραγματευόμαστε την δεύτερη διανιακή σύμβαση για την Ελλάδα και η Τρόικα βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις ημέρες και υπάρχει επίσης διαπραγματεύσεις με τον ιδιωτικό τομέα για να εξασφαλίσουμε τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, το PSI, την εμπλοκή, την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα που θα μειώσει την επιβάρυνση, το βάρος, το δανειακό της Ελλάδας με ε, στόχο να γίνει το δάνειο βιώσιμο, το χρέος βιώσιμο και να έχουμε ε, το 2020 μείωση κατά 120 δις έχουμε 130 δισεκατομμύρια για το, τη δεύτερη δανειακή σύμβαση. Μετά υπάρχει η Ιρλανδία. Εδώ η οικονομική βοήθεια βάση της σύμβασης είναι 85 δισεκατομμύρια. Η σύμβαση εφαρμόζεται τώρα με αρκετή επιτυχία. Δύσκολες αποφάσεις έχουν ληφθεί. Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν σκληρές αποφάσεις και οι αγορές καταλαβαίνουν ότι η Ιρλανδική κατάσταση αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Η τρίτη δανειακή σύμβαση αφορά την Πορτογαλία. Η οικονομική βοήθεια συμφωνήθηκε τον Απρίλιο 2011 για ένα σύνολο 78 δισεκατομμυρίων. Εδώ είναι πιο εύκολο, εν τρίτο, εν τρίτο, εν τρίτο, εν τρίτον η FSF, εν τρίτο η FSM και εν τρίτον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σύγκριση με την Ιρλανδία. Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μεγαλύτερες προκλήσεις και βεβαίως κάποια πρόοδος σημαντική έχει επιτευχθεί, αλλά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες και προβλέπεται ότι η οικονομική δραστηριότητα θα συμπεριστεί το 2012 πολύ περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά στα πλαίσια της σύμβασης και θα είναι ουσιαστικό η Πορτογαλία να υλοποιήσει πλήρως το πρόγραμμα, όχι μόνο το δημοσιονομικό σκέλος, την μείωση των δαπανών, αλλά επίσης και τις μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Εδώ βρισκόμαστε ως προς την υλοποίηση των συμβάσεων και των προγραμμάτων. Ξέρετε ότι υπήρξε συζήτηση χθες στο Συμβούλιο σχετικά με μια συμφωνία για το ESM. Υπάρχει μια οριστικοποίηση που περιμένουμε ε, του συμφώνου του δημοσιονομικού που ε, θα επιφέρει κάποια ε, πειθαρχία, έναν πόλο πειθαρχία που θα συνοδεύει τον πόλο αλληλεγγύης και όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα συνεκτικό σύστημα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ε, το ESM έχει συνολικούς πόρους της τάξης των 500 δισεκατομμυρίων και υπάρχει μια ρήτρα επισκόπησης τον Μάρτιο για να εξεταστεί η επάρκεια των πόρων. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είναι πυκνογραμμένες οι σημειώσεις σας, αλλά θα μπορούσατε να μας δώσετε μία σε έντυπη μορφή της παρεμβάσης σας στην γραμματεία, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε και να επωφεληθούμε. Έχουν ζητήσει αρκετοί το λόγο. Και εγώ θα ξεκινήσω με μια ερώτηση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε κάπως καλύτερα μαζί σας, κύριε Μπούτη. Το, το ποιο ταμείο θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά. Στην περίπτωση Πορτογαλίας ήταν ένα τρίτο, ένα τρίτο και ένα τρίτο. Μηχανισμός, μέσο και ε, δέλτα νιτάφ. Μας είπατε ότι ο μηχανισμός όχι μόνο έχει αναλάβει, αλλά έχει ήδη χορηγήσει 8 περίπου δις και έχει 48 υπογράψει ήδη ότι θα διανύμει στο μέλλον. Μέχρι τώρα λοιπόν έχετε δώσει 18 δις και άλλα 15 με 16 θα δώσετε σύντομα. Φαίνεται ότι υπάρχει εδώ ένα pattern, μια διαδικασία. Πρώτα χρησιμοποιείτε τον μηχανισμό που στηρίζεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και μετά περνάτε στο μέσο. Ίσως να είναι ευκολότερο να χρησιμοποιείτε πρώτα τον μηχανισμό σε σχέση με την ταχύτητα και την πρακτικότητα των παρεμβάσεων, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την χρήση αυτών των μέσων, γιατί το EFSM, ο Μηχανισμός Σταθεροποίησης, καλύπτει το σύνολο της Ένωσης και όχι μόνο την Ευρωζώνη. Αν υπάρξει λοιπόν μια χώρα εκτός Ευρωζώνης που αντιμετωπίζει δυσκολίες, δεν περισσεύουν και πάρα πολλά στα πλαίσια του EFSM. Βέβαια μπορείτε να περάσετε στην, στο μέσο της... Quite Well, those are my questions. Um, I'll go now to στο μέσο που προέρχεται από τη διαδικασία ελέγχου του ισοζυγίου πληρωμών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω πάρα πολλούς εγγεγραμμένους εδώ για να θέσουν ερωτήσεις. Roberto and Marianne Harkin. Θα ξεκινήσω με τρεις ερωτήσεις ε, κάθε φορά. Δεν μπορούμε να απαντάμε σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά, αλλά ας ξεκινήσει ο Σβέν και θα ακολουθήσουν άλλες δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την οργάνωση αυτής της ακροάσεως, αυτής της συνάντησης. Ήταν μια καλή ιδέα και δική σας και των συντονιστών. Μία ερώτηση θα ήθελα να θέσω. Όταν βλέπω τα διαφορετικά προγράμματα, και όταν βλέπω τους υπολογισμούς οι οποίοι μόλις δημοσιεύθηκαν σήμερα από το Ινστιτούτο Διεθνούς Οικονομίας του Κιέλου, το οποίο γνωρίζει ο κύριος Ρέγκλιν σαν Γερμανός, έχουν υπολογίσει ότι για τις διάφορες χώρες που υφίστανται κρίσεις ότι το απαραίτητο πλεόνασμα για τους προϋπολογισμούς τους αν θέλουν να εκπληρώσουν τους νόμους που έχουν ψηφιστεί στα πλαίσια του ΣΥΚΣΠΑΚ, δεν αναφέρομαι στο, χρηματο, στο δημοσιονομικό κομμάτι, αναφέρομαι σε αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο κοινοτικό. Λέγουν ότι για την Πορτογαλία, σαν παράδειγμα, αν ο ρυθμός ανάπτυξης επανέλθει στο 4%, που είναι βέβαια πάρα πολύ αισιόδοξο, πάντα θα απαιτείται ένα πλεόνασμα 9,2% στην περίπτωση της Ιρλανδίας 5,1%. Πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Εφόσον επανέλθει ο ρυθμός ανάπτυξης στο 4%. Για την Ελλάδα 27,8% πρωτογενές πλεόνασμα του ΕΠ έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι προβλέψεις που έχουν ήδη ψηφιστεί αυτό το Ινστιτούτο είναι ένα από τα πιο γνωστά ερευνητικά Ινστιτούτα στη Γερμανία και μόλις δημοσίευσε αυτές τις προβλέψεις. Μπορείτε να τα διαβάσετε στην ιστοσελίδα τους, δημοσιεύθηκε χθε και στο Spiegel. Αυτά τι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι οι χώρες αυτές, ακόμα και αν κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε, και το κάνετε αυτό, ακόμα και αν ηγηθείτε της εφαρμογής των προγραμμάτων, οι χώρες αυτές κάτω από τις παρούτες, παρούσες συνθήκες και με τις διαφορές στα επιτόκια που υπάρχουν, να ε, αποπληρώσουν τα χρέη τους. Οι χώρες αυτές χρειάζονται ισχυρότερα μέτρα από αυτά τα οποία έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στα πλαίσια των συμφωνημένων προγραμμάτων. Ποια είναι η ερώτησή μου λοιπόν. Πιστεύετε ότι τα προγράμματα μπορούν να πετύχουν, να φέρουν τις χώρες αυτές σε μια κάποια ισορροπία όταν υπάρχουν τόσο αρνητικοί δείκτες. Έχω και άλλους υπολογισμούς που έχουν γίνει στα πλαίσια του EFC, που δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τα προγράμματα τα συμφωνημένα. Οι λαοί υποφέρουν και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία, αυξάνεται η φτώχεια, αυξάνεται η ανεργία και αναρωτιέμαι αν έχει νόημα να πιέζεται τόσο πολύ κοινωνικά ο κόσμος, να πιέζεται τόσο πολύ και τόσο άδικα στα πλαίσια προγραμμάτων, τα οποία οικονομικά φαίνεται ότι δεν θα λειτουργήσουν. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Και μία τελευταία φράση. Ποτέ δεν υπήρξε μία χώρα του ΟΣΑ η οποία να έχει 5% πλεόνασμα του προϋπολογισμού για περίοδο άνω του ενός έτους. Και αυτό γιατί αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για τις οικονομίες των χωρών αυτών. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτό το οποίο ζητάμε σήμερα, απαιτούμε σήμερα από τις χώρες αυτές, είναι απαράδεκτο. Δεν θα πρέπει να μειωθεί το χρέος μόνο από, το τρέχον, ε, ε, από τα τρέχοντα έσοδα, αλλά και από συμπληρωματικά επιπλέον μέτρα. Υπάρχουν πολλές επιλογές εδώ. Αλλά δυστυχώς στις χώρες αυτές υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε τα επιβαρύνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η γραμματεία μου υπενθυμίζει ότι ένα λεπτό κάθε παρεμβαίνον πρέπει να έχει στη διάθεσή του. Καλώς το αναλώσατε εσείς τον χρόνο, τον χρόνο σας, γιατί ήταν σημαντικό αυτό. Το υπενθυμίζω λοιπόν. Τα ίδια αναφέρονται σε σχέση με τα στοιχεία αυτά. Ο επόμενος είναι ο Βουλφ Κλίντς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία σύντομη εκπροημή παρατήρηση. Ως Ευρωβουλευτής είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης ακριβώς εκείνα τα μέσα χρησιμοποιούμε που μετά την κατάρρευση των ε, Lehman Brothers οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση δηλαδή σε σχέση με την μόχλευση των ε, οικονομικών προϊόντων. Η ερώτησή μου, δεν περνάει ούτε μια εβδομάδα χωρίς κάποιος υψηλός αξιωματούχος, ο Μάριο Ντράγκη τώρα, και ο Ιταλός Πρόεδρος, Πρωθυπουργός διορθώνει ο μιλητής, να μην έχουν ζητήσει το EFSF ή το ESM να αυξηθεί στον χρηματοοικονομικό όγκο. Ερώτηση. Είπατε ότι κατά την άνοιξη θα επανεξεταστεί αυτό. Διερωτώ με, αυτό το θέμα δεν πρέπει να συνδυαστεί με αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να απαντηθεί σε σχέση με τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μισό δισεκατομμύριο, 500 εκατομμύρια ευρώ διέθεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις τάλες τράπεζες για να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο και δεν είναι και το τέρμα του προγράμματος. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας γι' αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Πώς τοποθετήσετε το ότι το, ε, έχουμε τώρα ε, την συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Έχει πραγματογνωμοσύνη, μπορεί να διατυπώνει σκληρές προτάσεις, το έχουμε συνηθίσει αυτό αλλά και ο Ζαν Πολτρισέ και ο Ντράγκη ε, ήταν εναντίον του, της συμμετοχής αυτής. Ουσιαστικά η Ευρωζώνη τα 330 δισεκατομμύρια, δηλαδή τόσους έχει πολίτες και, έχουν πολίτες και είπα πάνω 300 εκατομμύρια, να δούμε τι με τα 300 δισεκατομμύρια μπορεί να γίνει, 330 δισεκατομμύρια. Για την Ευρωζώνη και την υποβάθμιση της από τις, ε, τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, ακόμα δεν έχουν υπάρξει αρνητικές επιπτώσεις. Αλλά πώς το βλέπετε αυτό σε σχέση με το EFSF και το ESM και σε σχέση με αυτά που είπε ο Σβέν τελευταία, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε μια κατάσταση που είναι εξόφθαλμα σαφής. Όχι μόνο η Ελλάδα δεν έχει ρευστότητα, αλλά βρίσκεται στη γωνιά, στο περιθώριο και δεν έχει καν δυνατότητα να πληρώνει τους ε, μισθούς και τις συντάξεις. Ε, βρίσκεται πρώτης πτώχευσης. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε όπως μέχρι σήμερα. Πρέπει να σκεφτούμε αν εκ βάθρων χρειάζεται μια νέα προσέγγιση. Απόλυτα νέα. Ευχαριστώ. Σκληρά τα στοιχεία αυτά. Αν θέλετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις, στις απαντήσεις σας, να είσαστε σύντομοι. Γιατί έχουμε άλλους τρεις γύρους ερωτήσεων για την επόμενη μισή ώρα. Ο κύριος, όχι, ο κύριος Ρέγκλινγκ πρώτος. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε τις ερωτήσεις. Ο Μάρκο θα πάρει τις δύσκολες, εγώ τις εύκολες για να απαντήσω. Για την παρέμβασή σας, ε, όπως τοποθετηθήκατε, νομίζω μπορώ να απαντήσω. Ο, ε, επιμερισμός μεταξύ EFSF και του ESM έχει δύο τμήματα. Όταν αρχικά είχε αποφασιστεί ε, για μια περίοδο τριών ετών, για την Ιρλανδία τρία χρόνια, τριετής περίοδος, για την Πορτογαλία σχεδιάστηκε από την Ευρωζώνη, από την Ευρωομάδα πώς θα έπρεπε να ε, μοιραστεί αυτό και έτσι να δράσουμε. Τώρα η παρατήρηση βέβαια είναι σωστή που αναφέρατε ότι κατά τους πρώτους 12 μήνες έκανε περισσότερο το ESM από ότι το EFSF αλλά συνδέεται με πραγματιστικούς ρεαλιστικού λόγους και όχι για αυτού που υποθέτετε εσείς. Περνώντας από το EFSF1 στο EFSF2 θα ήταν πιο αποτελεσματικό να περιμέναμε και να μην χρησιμοποιούσαμε υπερβολικά το EFSF1, να αναμείνουμε με ότου θα ήταν λειτουργικό το EFSF2, διότι υπό το EFSF2 δεν θα χρειάζεται πλέον ε, η άμεση διάθεση των γρευτών όπως των μετρητών όπως στο EFSF1 λόγω των εγγυήσεων που έχουμε υπό το EFSF2. Είναι φθηνότερο δηλαδή υπό το πλαίσιο του EFSF τώρα πλέον εφ' αυτό το οποίο μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει υπό το EFSF1. Ή θα είχε νόημα λοιπόν να μην χρησιμοποιήσουμε υπερβολικά το EFSF1, να ζητήσουμε το ESM να εμπλακεί περισσότερο, να γεφυροποιήσει αυτή την περίοδο και μετά από μια περίοδο τριών τριών ετών θα είχαμε ακριβώς τα αριθμητικά μεγέθη που είχαν συμφωνηθεί κατά την έναρξη του προγράμματος. Στον κύριο Κλίντς, θα ήθελα να πω να μην συγκρίνουμε αυτά τα οποία κάνουμε στο EFSF και σε σχέση με το ESM με μοχλικά προϊόντα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν και που οδήγησαν στην κρίση της αγοράς των αγορών ξεκινώντας με την αγορά στέγης στη ΣΥΠΑ με τη φούσκα των στεγαστικών δανείων. Αυτά που κάνουμε είναι διαφανή. Θα το συνέκρινα αν κάποιος αγοράζει ένα διαμέρισμα ή ένα ε, σπίτι 20% δίνεται ως προκαταβολή και το υπόλοιπο 80% προσπαθείτε να το καλύψετε μέσω των τραπεζικών δανείων. Είναι μια απλή ε, διαδικασία που όλοι την κατανοούν και αυτό κάνουμε και εμείς τώρα. Προσπαθούμε να επανέλθουν οι ιδιωτικοί επενδυτές στην Ευρώπη για να αγοράσουν εκείνα τα ομόλογα που δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να αγοράσουν. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις νότιες, τις χώρες του νότου της Ευρώπης και φυσικά δεν μπορεί να συγκριθεί απόλυτα σε σχέση με την οικονομική κρίση το ένα με το άλλο ε, όσον αφορά αυτές τις διεργασίες Έχετε όμως δίκιο στο ότι η πρόβλεψη των δανείων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δραματικά αυξήθηκε το Δεκέμβριο σε σχέση με την διάθεση κονδυλίων για μια τριετή περίοδο που μπορεί να βοηθήσει, το βλέπουμε αυτό, το καθιστά ευκολότερο για τις τράπεζες να επαναγοράσουν κρατικά ομόλογα. Και έτσι θα δούμε σε ποιο βαθμό αυτό θα, γίνει, θα είναι εφικτό και θα συνεχιστεί. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που το 2010 είχε αναφερθεί ότι θα έπρεπε να εμπλακεί και εξεταζόταν η συμμετοχή του ή όχι. Τώρα σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά, βλέποντας ότι έχει διαδοθεί σε μεγάλο βαθμό η οχι τωρα σημερα σχεδον δυο χρονια μετα βλεποντα οτι εχει διαδοθει σε μεγαλο βαθμο η κριση και πλήττει διάφορε χώρε. βλέπουμε και ότι ο όγκο των κονδυλίων που χρειάζεται για να βοηθηθούν αυτέ οι χώρε είναι σημαντικά αυξημένο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία αυτή τη στιγμή ότι η εμπλοκή του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου είναι υποφελή όσον αφορά και κονδύλια και πραγματογνωμοσύνη που παρέχει. Και είμαι σίγουρο ότι ο κύριο Μάκο Μπούτι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου είναι πολύ καλή. Και όσον αφορά και το μέσο για τον ισοσκελισμό προπολογισμών και για τη βοήθεια χωρών εκτό ζώνη ευρώ, είναι και αυτό σημαντικό στοιχείο τελική μου παρατήρηση για την υποβάθμιση του EFSF που έγινε πριν την προηγούμενη Δευτέρα από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Είχαμε προηγούμενα και την υποβάθμιση κάποιων χωρών στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση από τους οίκους αξιολόγησης. Και βλέπουμε τώρα αυτή την υποβάθμιση. Δεν είναι εκπληκτικό ότι κατά μία κλίμακα υποβαθμίστηκε αυτό το μέσο. άλλες, οι άλλοι οίκοι ε, Moody's ε, και ε, δεν το, δεν το έκαναν αυτό. Είπαν ότι δεν είχαν την πρόθεση σε σχέση με την υποβάθμιση της Γαλλίας. Από πλευράς του άλλου οίκου όμως έγινε αυτό. Έχουμε λοιπόν αυτό η προσέγγιση. Αυτή τη στιγμή ένας οίκο από τους τρει το έκανε αυτό και μόνο για μακροπρόθεσμες προοπτικές, ε, για τις ε, μέσοπρόθεσμες, υπάρχει πρόθεσμες προοπτικές ε, επιστοληπτικής αξιολόγησης έχουν ακόμα την ανώτατη βαθμολογία και αυτό δεν πρέπει λοιπόν τώρα να μας παραξενεύει. Ακόμα και μετά την υποβάθμιση προσφύγαμε στι αγορές και καλύψαμε υπερακούντος τις ανάγκες μα. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει, να μας παξενεύει αυτό. Όταν το EFSF θα είναι λειτουργικό, μετά από πέντε μήνες θα είναι πολύ λιγότερο ευπρόσβητο το ε, ESM σε τέτοιου είδους ε, διαδικασίες. Θα λάβει τον λόγο ο Μάρκο τώρα. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα ερώτηση και ε, πρέπει να προκαλέσει αρκετές δυνατότητες να απαντηθούν αυτά τα θέματα. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην αρχή χρησιμοποίησαμε περισσότερο την δυνατότητα που είχαμε ε, για τις υποδομές που είχαμε στη διάθεσή μας ε, και μετά από τις ε, διεργασίες της Συμφωνίας της Βασιλείας είμαστε πιο έτοιμοι από το EFSF να ξεκινήσουμε να δρούμε με το ESM και έτσι επιλέξαμε να περάσουμε με αυτόν τον τρόπο στις αγορές για να καλύψουμε τις ανάγκες μας όσον αφορά τη σύγκριση με το EFSF. Τώρα όλες οι μελέτες όσον αφορά την μελέτη που αναφέρατε δεν την γνωρίζω, δεν μπορώ να σχολιάσω λοιπόν όσον αφορά τα πορίσματα αυτής της μελέτης. Αν όμως τα αριθμητικά μεγέθη είναι αυτά τα οποία αναφέρατε, δεν ξέρω αν πρέπει και αξίζει να μελετηθεί αυτό σε βάθος, διότι αν αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή διαφορά μεταξύ των επιτοκίων σε σχέση με την σταθεροποίηση του χρέους είναι σαφές ότι χρειάζονται τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα. Έτσι δεν είναι για την Ελλάδα ένα πρωτογενές πλεόνασμα 25% του ΑΕΠ. Ανήκουστο αυτό αν εγώ ή κάποιο συνεργάτη μου το ε, κατέγραφε αυτό σε ένα σημείωμα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να προβιβαστεί τους τα επόμενα δέκα έτη να ε, προαχθεί βαθμολογικά στη σταδιοδρομία του. Σαφώ αυτό που έχουμε τώρα για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα επιτόχια και τα spreads, γι' αυτό ελήφθη η απόφαση με τα προγράμματα αυτά να βοηθηθούν οι χώρες αυτές να ε, τεθούν εκτός αγοράς και εμείς να δράσουμε. Βρισκόμαστε στην διαδικασία εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων ακριβώς, υποστήριξης, διάσωσης αυτών των χωρών. Και παρότι φυσικά θα είναι πολύ επώδυνες οι επιλογές που θα πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο, στο πολιτικό εθνικό επίπεδο, πιστεύουμε ότι θα στεφθεί με επιτυχία με το εγχείρημα αυτό. Τώρα τα ίδια τα αριθμητικά μεγέθη. Δεν μου φαίνεται ότι είναι ορθά 5% πρωτογενές πλεόνασμα όπως αναφέρθηκε για ένα χρόνο μόνο, μόνο ετός. Ε, τώρα σε σχέση με την πείρα, την ε, ε, εμπειρία στην Ευρώπη έχουμε την περίπτωση του Βελγίου παράδειγμα. Επίσης και της Ιταλίας που διατήρησαν ένα πρωτογενές πλεόνασμα 5,5% για κάποια αρκετά χρόνια και μπόρεσαν να μειώσουν ε, το φάσμα της ε, κρίσης όσον αφορά το χρέος που έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα. Τώρα, αυτό σε σχέση με την Ιταλία, υπό τη δέσμευση του τότε, του τότε Πρωθυπουργού Τσάμπη για την προσχώρηση, την ένταξη στη ζώνη ευρώ και για το Βέλγιο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν είχε 135% ε, χρέος του ΑΕΠ το Βέλγιο και κατόρθωσε να το μειώσει σε ένα 85% του ΑΕΠ. Τώρα, για την Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση και γι' αυτό γνωρίζουμε και γι' αυτό τον λόγο βρισκόμαστε σε επαφή με τον ιδιωτικό τομέα, με τους ιδιώτες, για να μειωθεί ο όγκος του χρέους μέσω κουρέματος, κουρέματος 50% που αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως τμήμα του δεύτερου προγράμματος θα, υπάρξει, θα υπάρξουν 30 δισεκατομμύρια για να βοηθηθεί αυτός ο στόχος και ο στόχος θα είναι να μειωθεί το χρέος της Ελλάδας η υπερχρέωσή της στο 120% του ΑΕΠ το 2020 και κάτω από το 100% του ΑΕΠ μέχρι το 2030 και για την περίπτωση της Ελλάδας αυτό σε συνδυασμό με το δεύτερο ε, πρόγραμμα το οποίο ε, σίγουρα θα είναι ένα πολύ επώδυνο πρόγραμμα με πολύ οδυνηρές επιπτώσεις θα καταφέρουμε να φέρουμε το χρέος σε κάποιο βιώσιμο επίπεδο. Τώρα, σε όλες αυτές τις χώρες, από την άλλη πλευρά, Ιρλανδία, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των διαθωτικών μεταβολών, διαθωτικών αλλαγών. Δεν υπάρχει τρόπος να διατηρηθούν τα δημοσιονομικά με υγιή βιώσιμο τρόπο αν δεν έχουμε υγιή ανάπτυξη μέσω διαθωτικών αλλαγών. Όλα αυτά καταλήγουν στο τέλος τέλος ε, στο να τεθεί έμφαση, με ιδιαίτερη έμφαση, ο τόνος στις διαθροτικές ε, αλλαγές. Και πρέπει να πω ότι σε όλες αυτές τις χώρες ε, λαμβάνουμε υπόψη ε, ε, τον ισοδίκαιο τρόπο δράσης και εφαρμογής όσον αφορά την αντιμετώπιση του χρέους. Είναι ένας περιορισμός βέβαια αυτός που έχουμε στη δράση μας και προσπαθούμε να προστατέψουμε τα χαμηλά εισοδήματα, τους πιο φτωχούς ε, στην κάθε χώρα από ιδιαίτερα υπόδεινα πλήγματα. Βλέπω τώρα ότι η πρόεδρος όμως ανησυχεί επειδή μακρηγόρησα. Πράγματι ανησυχώ, διότι πρέπει τέσσερις ακόμα ερωτήσεις να παίρνουμε ταυτόχρονα και πρέπει να ολοκληρώνουμε κάθε γύρω Δέκα λεπτά. Εντάξει, τέσσερις ερωτήσεις και δύο απαντήσεις, Δέκα λεπτά συνολικά. Ε, κάντε τον υπολογισμό, δείτε τι πρέπει να κάνουμε για να το καταφέρουμε. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση Πρόεδρε, βλέπω ότι η συζήτηση, η συζήτηση είναι τόσο ενδιαφέρουσα ότι πρέπει να συνεχιστεί αν σήμερα δεν μπορέσει να ολοκληρωθεί. Πρέπει κάποτε να συνεχιστεί γιατί είναι πολύ σημαντικά τα θέματα. Ερωτώ τον κύριο Ρέγκλινγκ πρώτα καταρχήν. Μπορώ να φανταστώ βέβαια μόνο κύριε Ρέγκλινγκ, εδώ είμαι, εδώ βρίσκομαι. Μπορώ να φανταστώ ότι εσείς ε, έχετε ενεργοποιήσει ένα διακυβερνητικό όργανο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα κοινοτικό μέσο να λειτουργήσει πόσο υψηλό είναι το κόστος ότι δεν έχουμε ένα διακοινωτικό μέσο το οποίο ε, ενεργοποιούμε αλλά μόνο ένα διακυβερνητικό μέσο. Δεν είναι ακαδημαϊκό το ερώτημα, δεν είναι θεωρητικό. Αν τα πράγματα πάνε στραβά ποιος θα είναι υπεύθυνο στο τέλος τέλος διότι εδώ διαθέτουμε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθενται και κονδύλια του Κοινοβουλίου. Αν δεν γνωρίζετε τα μεγέθη, τα αριθμητικά μεγέθη του Ιδρύματος Οικονομικών Μελετών του, Κι, του Κιέλου, στο Κιρ της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Πείτε μας ποια είναι τα δικά σας αριθμητικά μεγέθη. Υπό ποιου όρους, με ποιο τρόπο θα αναπτυχθούν αυτές οι χώρες και πώς θα εξελιχθούν. Διότι με δίκαιο, ε, είναι δίκαιο να λέμε πολλοί από εμά ότι δεν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και καμιά ιδέα για την οικονομική ανάπτυξη με όλα αυτά τα μέτρα. Αντίθετα υπάρχει ο κίνδυνος που ελοχεύει να καταλήξουμε σε μια καταστροφή της ανάπτυξης και του αναπτυξιακού προγράμματος είναι όλα αυτά, αλλά πότε θα αποδώσουν καρπούς, πότε θα έχουμε τον πυρήνα των καρπών αυτών των προτάσεων και τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά δεν μπορούν ε, να επιτευχθούν αυτή τη στιγμή. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε οι αναπτυξιακές δυνάμεις σε αυτές τις κοινωνίες να μπορέσουν να τονωθούν. Παράδειγμα, σαν με το πρόγραμμα Marshall μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σχέδιο Marshall. Ευχαριστώ. Ε, είναι ε, ερώτηση ενός μάνατζερ ε, που ακούει αυτό που θέλει να ακούσει και όχι την πραγματικότητα. Θα σας στείλω τα έγγραφα του ΟΣΑ, τα έγγραφα του ΑΕΦΟ. Η ΑΕΦΟ μας λέει ότι το Ινστιτούτο του Κι λέει ότι αυτό που χρειάζεται στην Πορτογαλία με, με υπόθεση 2% ε, και 6% πρωτογενή ε, πλεόνασμα. Ενώ η Ελλάδα χρειάζεται για το ίδιο σενάριο 22%. Ίσως δεν σας αρέσουν αυτοί οι αριθμοί, αλλά είναι η πραγματικότητα. Αυτό περιλαμβάνει την υπόθεση ότι το spread θα μειωθεί κατά το ίμιση η διαφορά επικοτοκίων με τη Γερμανία. Μπορεί να μην σα αρέσουν οι αριθμοί αυτοί, αλλά υπάρχουν οι αριθμοί αυτοί. Μπορεί να επικρίνετε του οικονομολόγους, αλλά θα πρέπει και τα, τα δικά σα. Βρισκόμαστε σε μια μη βιώσιμη κατάσταση αυτή τη χώρα και όχι μόνο στην Ελλάδα και κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Για πάνω από ένα χρόνο η Κομοσιό είπε ότι δεν θα υπάρξει αναδιόρθρωση του ελληνικού χρέου. Ήταν η ιδεολογική αυτή στάση, μετά αναγνωρίσατε ότι σφάλεται. Έχω ερωτήσεις για τον κύριο Ρέγκλινγκ. Ε, ποια θα είναι τα υπέρ και τα ε, κατά σχετικά με τις άδειες της ε, τραπεζικές. Αυτή η υπόθεση έχει διατυπωθεί από ορισμένη και από την κόμμα μου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, ερώτηση και στους δύο σας. Αν φανταστούμε ότι υπάρχει χρεοκοπία της Γρέσης της Ελλάδας και η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει, δεν βλέπω να μπορεί να αναστηθεί, ε, τι, μέσα θα έχει το EFSF και η e FSM σε τέτοια περίπτωση. Ποια θα είναι η προτεραιότητα για τα υπόλοιπα ε, κονδύλια που μπορούν να μοχλευθούν από τις δύο οργανώσεις σας σε μια τέτοια περίπτωση. Και τελευταία ερώτηση στον κύριο Μπούτη. Λέτε ότι ε, λαμβάνετε υπόψη την δικαιοσύνη, την ισότητα ποια είναι τα πρακτικά μέτρα που δείχνεται ότι όντως η Επιτροπή έχει λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των πιο ε, ευάλωτων στρωμάτων της κοινωνίας. Ευχαριστώ, Έτη. Άντολιν πρώτον. Ο ναι. Αντολίν, ευχαριστώ πολύ. Ετέθησαν ήδη ερωτήματα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θα ήθελα να μας εξηγήσετε το Ευρωπαϊκό Μέσο της Οικονομικής Σταθεροποίησης που έχει δύο νέα έργα παρέμβαση στις δευτερογενείς αγορές και την επανακεφαλαιοποίηση. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το νόημα των παρεμβάσεων αυτών ιδιαίτερα στη δευτερογενή αγορά. Ποιε είναι οι σχέσεις ο συσχετισμός με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την άλλη πλευρά για το EFSM Πρόκειται εδώ για ένα μέρο το οποίο χρηματοδοτείται από του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιονομικά. Θέλω να ξέρω τι γίνεται σε σχέση με τον στο συσχετισμό με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την πληροφόρηση και ενημέρωση και που κυρίω οι και προποθέσει ε, πρέπει να λειτουργεί. Ετέθη αυτέ τι μέρε ε, ένα θέμα για τον όγκο, των χρηματοοικονομικών, των ποσών που θα πρέπει να διατίθεται. Ποιο είναι, ποια είναι η δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή λαμβάνοντας υπόψη την πιστοληπτική υποβάθμιση που είχαμε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε και με τις υπόλοιπες ερωτήσεις γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να τις ακούσουμε καν. Η Ελίζα, επόμενη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Εδώ βρίσκομαι εγώ. Σας ευχαριστούμε που παρίσταστε. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω να ανασκοπήσετε προς το παρελθόν και να αξιολογήσετε, να σταθμίσετε την εξέλιξη την οποία βιώσαμε και το τι συνέβη. Και για την αμφισβήτηση των αριθμητικών μεγεθών για, όπως παρουσιάστηκαν από τους προηγούμενους αγορητές. Ακόμα και αν δεν έχετε στη διάθεσή σας αυτά τα αριθμητικά μεγέθη, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι το κόστος του δανείου σε χώρες όπως ιδιαίτερα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα και στην Πορτογαλία και η χρονική περίοδο σε σχέση από κοινού με τα μέσα που προτάθηκαν ή επιβλήθηκαν κιόλα. Δεν μπορούσαν όλα αυτά να λειτουργήσουν. Ω οικονομολόγο μπορούσε κανεί να το δει αυτό. Ποτέ δεν θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικά και αυτό είναι η πραγματικότητα. Και επιπλέον ποτέ δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν με κανέναν και σε κανένα. Φυσικά κάνετε λόγο για διαθροτικέ μεταρρυθμίσει. Οι διαθροτικέ μεταρρυθμίσει όμω παίρνουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μεταφραστούν σε ανταγωνιστικότητα μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα έχουμε παντού ύφεση. Έχουμε τα εξαπλά μέτρα, το six pack, ελπίζοντας ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την ίδια την ανάπτυξη. Δεν έγιναν όλα αυτά. Και τώρα έχουμε περιοριστική και νέες περιοριστικές διαστάσεις ε, του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Πάλι ε, επιβάλλοντας πίεση για βραχυπρόθεσμες προσαρμογές με βάση μια δισκαμψία και μια επιβολή περιορισμών για την αντιμετώπιση λέει, των ελλημάτων και του χρέους. Είναι αυτή η χρονική στιγμή για να γίνουν αυτά. Αυξάνονται τα spread. Ε, δεν λειτουργούν όλα αυτά τα μέσα και οι ρήτρε ασφάλεια. Οι συστάσει δεν λειτουργούν σωστά. Τώρα είναι η χρονική στιγμή για να περάσουμε εκτό αυτού του στενού πλαισίου και να μην στριφογυρίζουμε σε ένα φαύλο κύκλο γύρω από προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Το θέτω ομά υπάρχει αιμονή και επιμονή σε συστάσεις που ποτέ δεν μπορούν να είναι ρεαλιστικές και αποτελεσματικές. Εδώ λείπει το στοιχείο της ανάπτυξης και το στοιχείο της απασχόλησης. Ζητείτε από χώρες να πιεστούν, να στραγγιστούν για να υπάρξει λέει αυτή η ανάκαμψη. Έχει συρρυκνωθεί η συνιστόσα της ανάπτυξης. Είναι μια σπυροειδής ε, εξέλιξη προς την ύφεση και τον μαρασμό και δεν υπάρχει διέξοδος από αυτό Πρότασή μου είναι να προχωρήσουμε με τελείως διαφορετικά μέτρα, με τελείως διαφορετικά πολιτικά και οικονομικά κίνητρα για να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε τα κοινά προβλήματά μας. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Φοβούμαι ότι υπάρχει μόλυνση και επιμόλυνση με αυτή την ύφεση και την ε, διάλυση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτά τα περιοριστικά μέσα καταστολής πανευρωπαϊκά και στη ζώνη ευρώ. Λυπούμε, αλλά δεν μπορούσα να απόσχω, έπρεπε να τα πω αυτά σε Ευχαριστώ. πολύ. Ίσως θα έπρεπε να είναι κάποιοι άλλοι ε, για να τους κάνετε αυτές τις ερωτήσεις, να πυροβολήσετε με αυτές τις ερωτήσεις. Θα έχουμε 10 λεπτά επιπλέον από πλευράς διαμηνίας, αλλιώς θα πρέπει να συνεχίσετε στα αγγλικά. Συνεχίζω σε αυτά τα οποία έλεγε μόλις προηγουμένως τη Ελίζα. Όταν βλέπει κανείς τους οικονομολόγους από κοντά, διερωτάτε αν υπάρχουν πραγματικά σήμερα αποδείξεις για κάποιες ε, διευρυντικές θα έλεγα επιπτώσεις της οικονομικής βοήθειας την οποία δίνουμε μέσω του EFSF και του EFSM. Σχετικά με το PSI στο οποίο αναφερθήκατε μόνο τροχάδι, μπορείτε να μας πείτε τι βλέπετε σε σχέση με τον χρονισμό και την πιθανότητα ε, χρήσης των CDS Muito, muito obrigado. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα δύο ερωτήσεις να διατυπώσω άμεσες σε σχέση με τις ανησυχίες που προαναφέρθηκαν από άλλους συναδέρφους ε, ε, όπως από την κυρία Λίζα Φερέδα. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς την δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι στο μέλλον πλέον ο επενδυτής ο επενδυτής της προσφυγής που θα δρούσε. Και επίσης, κατά δεύτερο λόγο, μια και μιλάμε για κρατική υπερχρέωση και την αντιμετώπιση του κρατικού χρέους, πώς αναλύετε εσείς μια πρόταση που έγινε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, τους German wise men, τους Γερμανούς σοφούς όπως τους αποκαλούμε, που προτείνουν την ύπαρξη ενός ταμείου για να αγοράσει αυτό το ταμείο το χρέος το οποίο θα είναι ε, πάνω από το 70%. Ένα ταμείο διάσωσης δηλαδή με άλλα λόγια για μια παρατεταμένη περίοδο. Πώς αναλύετε και αντιμετωπίζετε εσείς ακριβώς αυτήν την πρόταση. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Λία. Ευχαριστώ ε, που ήρθατε εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο διότι οι πληροφορίες που έχουμε στον τύπο είναι αδιαφανείς. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τη λειτουργία του επομένου μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Σταθερότητας. Ποιος θα εγγυάται για αυτόν τον μηχανισμό, δεν μας λένε. Μας λένε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά αυτός είναι 140 δισεκατομμύρια και έχει ήδη διατεθεί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τον εγγυάται τον μηχανισμό ή κάτι άλλο. Και ε, ποιοι θα είναι οι τίτλοι που θα εκδοθούν από αυτόν τον μηχανισμό, διότι θα πρέπει να συλλέξει κονδύλια, κεφάλαια στην αγορά. Θα είναι ευρωομόλογα και ίσως τότε αυτό θα πρέπει να προετοιμαστεί με κατάλληλο τρόπο, διότι ε, η λειτουργία του σημερινού EFSF είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Τα κρατημέλη δεν μπορούν να τον εγγυηθούν διότι υπάρχει κρίση δημοσίων οικονομικών. Έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εγγυηθεί αυτό το ταμείο και η μόχλευση για την οποία μιλήσατε είναι πάρα πολύ επικίνδυνη διότι είναι τίτλοποίηση χρεών επικινδύνων ε, για να μπορεί κανείς με παράγωγα προϊόντα να αποκτήσει κονδύλια, κεφάλαια, προϊόντα, ε, μια αποτεμίευση και τα προϊόντα αυτά το ξέρουμε. Ε, το, με τα subprimes είδαμε, με τα ενυπόθηκα επικίνδυνα στεγαστικά δάνεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά νομίζω μόλυναν τους ισολογισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ ανησυχώ, μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο. Ρομπέρτο. Ευχαριστώ. Δεν θα επανέλθω στους λόγους τους οποίους υπενθύμισε και ο Μπούρμαν, στους λόγους που περιορίζουν τον πιθανό αποτελεσματικό ρόλο του EFSF, του EFSM, ιδιαίτερα τον διακυβερνητικό χαρακτήρα του μέσου που δημιουργεί προβλήματα στη χρηματοδότηση. στη μεμονωμένη εθνική συμμετοχή, στην παροχή εγγυήσεων επίσης από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Θέλω και εγώ να στραφώ λίγο προς το μέλλον πάντως και να επανέλθω σε θέματα βέβαια τα οποία έχουν ήδη τεθεί. Για τις αλλαγές σε επίπεδο τραπεζικό. Ποιοι είναι οι λόγοι, αν υπάρχουν νομικοί, πολιτικοί λόγοι ή πολιτικές αξιολογήσεις που μέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί υπόψη. Τι είναι αυτό το οποίο θα επέτρεπε να υπάρξει επί τη βάση του 123.2 μια καλύτερη και διαφορετική σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα, για ερώτηση προς τον Μπούτη σχετικά με το ταμείο που κρατά το χρέος, που συλλέγει το χρέος. Ο μηχανισμός αυτός στην ουσία έχει τεθεί λίγο στο περιθώριο και δεν έχουμε πληροφορίες για, το, για τη νομική του βάση, σαν παράδειγμα. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό παραπέμπει η νομική αυτή βάση σε ισχύουσες συνθήκες, αντίθετα με το EFSF και τα άλλα ταμεία. Τρίτον, το EFSM τώρα, ο Κοινοτικός Μηχανισμός Σταθεροποίησης. Υπάρχει μια εκτίμηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομικές συνέπειες σε επίπεδο προϋπολογισμού, σε επίπεδο ιδίων πόρων και σε επίπεδο πιθανών πολιτικών μέσων έτσι ώστε να υπάρξει μια ισχυροποίηση επιτέλους του EFSM. Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, δύο προσκεκλημένους. Η Ιρλανδική κυβέρνηση αύριο θα δώσει 1,25 δις ε, στην Anglo-Irish Bank, που δεν υπάρχει ουσιαστικά, έχει πτωχεύσει η τράπεζα αυτή, είναι μια τράπεζα ζόμπι. Τον Μάρτιο 3,1 δις στην ίδια επίσης ε, τράπεζα και σε άλλους πιστωτές. Το κάνουμε αυτό γιατί στην ουσία δανειζόμαστε με επιτόκιο 8,6%. Το συνολικό κόστος για να διασώσουμε μία τράπεζα μόνο είναι 47 δις για μία τράπεζα, αλλά υπάρχουν και άλλες τράπεζες στη σειρά. Η πρώτη ερώτησή μου είναι η εξής λοιπόν. Πώς μπορεί να δικαιολογήσει κανείς για μια χώρα η οποία περνάει την διαδικασία που περνάμε εμείς, να πληρώνει αυτές τις απαράδεκτες, αυτά τα απαράδεκτα επίπεδα επιτοκίων. Μας είπατε ότι η διαδικασία στην Ευλανδία πηγαίνει καλά. Μακάρι να ίσχυε, μακάρι να μου έλεγαν οι συνάδελφοι στο διάδρομο ότι τα πράγματα πάνε καλά και να έλεγαν ναι. Όλοι θα θέλαμε κάτι τέτοιο, όλοι θα θέλαμε να πάνε καλά, αλλά δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Το χρέος αυξάνεται, το εισόδημα μειώνεται, δεν χρειάζεται να σας δώσω, αλλά η ελπίδα την οποία είχαμε είναι οι εξαγωγές και αυτοί μειώνονται τους τελευταίους πέντε μήνες. Είμαστε κάτω από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο ε, εξαγωγών. Μιλάμε τώρα για μία πορεία προς την ύφεση. Δεν ξέρω αν είμαστε στη μέση αυτής της πορείας. Δεν μπορείτε όμως να λέτε ότι η κατάσταση πηγαίνει καλά. Δεν πηγαίνει καλά η κατάσταση και ένα τελικό σχόλιο. Δεν είμαι μέλλον της Επιτροπής και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να πάρω το λόγο. Έχουμε έτσι και αλλιώ και το six-pack και το δημοσιονομικό πακέτο με συγκεκριμένους κανόνες. Αλλά ανάμεσα στο 2002 και το 2008 η Ιρλανδία έμεινε στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και πήγε πολύ καλύτερα από ότι η Γαλλία και η Γερμανία. Αλλά αυτό τελικά δεν μας έσωσε. Οπότε ναι, χρειάζεται σίγουρα να σεβαστούμε τους κανόνες τους δημοσιονομικούς. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει όμως και μια διαφορετική δυνατότητα ανάπτυξης και μια διαφορετικού τύπου διαγραφή χαριστική αν θέλετε χρέος. Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα χρεώσουμε τις επερχόμενες γενναίες για πολύ καιρό. Λοιπόν, ακούσαμε λόγια γεμάτα ειλικρίνεια από όλα τα μέλη εδώ. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά κοινά στοιχεία σε, αυτά τα οποία ακούσαμε και δεν είναι καθόλου ευχάριστα αυτά τα οποία ακούσαμε. Και θα θέλαμε από πλευρά σας κάποιες ειλικρινείς παρακαλώ απαντήσεις στο βαθμό του δυνατού και σε επίπεδο επιτοκίων είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει γιατί πολλές φορές ε, τα επιτόκια ήταν σε αγορευτικά επίπεδα, δεν έπρεπε να πάρουν χρήματα με τέτοια επίπεδα επιτοκίων. Γιατί έτσι κι αλλιώς ε, αυτά τα χρήματα δεν αρκούν για να σωθούν οι συγκεκριμένε χώρες. Δεν έχουμε πάνω από δέκα λεπτά, δεν ξέρω ποιος από τους δυο σας θα ξεκινήσει. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ευθέως σε σχέση με όλες αυτές ε, τις ερωτήσεις. Ακούσαμε ε, Ιρλανδικό μέλος του Ευρωκοινοβουλίου ε, στο Eurogroup μπορώ να σας πω και ο, στην Τρόικα πιστεύουν ότι το πρόγραμμα λειτουργεί καλά. Δεν λέμε ότι δεν υποφέρει ο πληθυσμός αλλά έχει αναδιαρθρωθεί ο τραπεζικός τομέας ε, το έλλειμμα τρεχουσών ε, συναλλαγών πέρσι έγινε πλεόνασμα και το πλεόνασμα αυξάνει και αυτή είναι ένδειξη ότι η ανταγωνιστικότητα αποκαθίσταται. Ξέρουμε από όλου τους δείκτε ότι η μισή ανταγωνιστικότητα που είχε χαθεί στην πρώτη ε, δεκαετία έχει ανακτηθεί στην Ιρλανδία. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίω δεν τελείωσε η διαδικασία, ότι τα μισά έχουν γίνει με μεγάλο άχθος ε, για, και οδύνη για τον πληθυσμό. Δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις. Η Ιρλανδία κάνει μεγάλη πρόοδο και δεν είναι σωστό, όπως λέτε, ε, να πείτε ότι οι αντιπυρικές ζώνες ε, δεν λειτουργούν καλά. Το επιτόκιο έχει μειωθεί κατά το ίμιση στην Ιρλανδία ήταν 14% ε, και τώρα είναι 7,5% για τα κρατικά ομόλογα. Περίπου έχει ε, κοπεί στη μέση το επιτόκιο, η απόδοση των ομολόγων. Είναι ένα γεγονό. Δεν μπορείτε να πείτε λοιπόν ότι παντού τα επιτόκια ανεβαίνουν. Όχι, όχι. Μειώθηκαν τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες. Αυτά για την ε, γενική εκτίμηση. Για το πιο συγκεκριμένο ερώτημα, κύριε Μπούλμαν, δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να πει ότι το κόστος οργάνωσης του EFSF με διακυβερνητικό τρόπο είναι υψηλότερος από ότι να οργανωθεί με κοινοτικό τρόπο, με την κοινοτική μέθοδο. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές ε, πολιτικά στοιχεία γύρω από όλα αυτά. Δεν ήταν η ερώτησή σας. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι, θα ήταν ψηλότερο το οικονομικό κόστος ε, την εποχή πριν από δύο χρόνια ο μόνος ταχύτερος, ταχύτατος τρόπος να γίνει αυτό, να δημιουργηθεί ήταν ο, ο διακυβερνητικός με βάση το δίκαιο του Λουξεμβούργου. Ήταν ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε γρήγορα το ESM. Θα είναι βάση του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς συνθήκης. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Αν το κάναμε αυτό με το EFSF δεν θα είχε λειτουργήσει μέσα σε λίγους μήνες. Και αυτό ήταν, γινόταν μόνο ε, με την προσέγγιση προσέγγιση και δεν νομίζω ότι το οικονομικό κόστος ήταν υψηλότερο. Ε, το θέμα από το EFSM ήρθε από πάρα πολλούς ε, ομιλητές, αν είναι της τελευταίας καταφυγής ε, δανειστής πολλά κράτη-μέλη πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει σαφής καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στη δημοσιονομική πολιτική και στη νομισματική πολιτική. Είναι μια καλή αρχή και αυτό εγγυάται την ανεξαρτησία κεντρικής τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι τελευταίας καταφύγης δανειστής για τις τράπεζες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, κυρίως τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά ε, η ΕΚΤ δεν είναι για τα κρατικά ομόλογα ο δανειστής τελευταίας καταφυγής. Και αυτό από νομικής απόψεως δεν γίνεται αν η FSF, η FSM ε, είχαν μια τραπεζική άδεια ε, θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν οι κυβερνήσεις διότι δεν επιτρέπεται από την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί ομιλητές επίσης είπαν ποια είναι η καλύτερη χρήση των πόρων που απομένουν του EFSF, ESM αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για παρεμβάσεις στη δευτερογενή αγορά, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες. Για την ώρα, εξετάζοντας μόνο το EFSF, έχουμε δεσμεύσει μόνο 10% της ικανότητας που έχουμε ε, για την Ιρλανδία και Πορτογαλία. Ε, χρειαζόμαστε μεγάλο κομμάτι δανεισμού για την Ελλάδα αλλά θα παραμείνουν αρκετά δισεκατομμύρια. Δεν ξέρουμε ποιοι θα χρειαστούν αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη χώρα που θα ζητήσει βοήθεια. Αυτό θα εξαρτηθεί. Πρώτο δεν ξέρουμε αν θα έρθει κάποια χώρα, αν έρθει κάποια χώρα θα εξαρτηθεί από το είδους των προβλημάτων που θα έχει χώρα αν είναι στον τραπεζικό τομέα. Ίσως θα πρέπει να γίνει ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών αν είναι χώρα που χρειάζεται ε, βοήθεια για την μείωση των επιτοκίων στη δευτερογενή αγορά. Θα έχουμε παρεμβάσει στη δευτερογενή αγορά. Όλα εξαρτώνται από τη χώρα που θα έρθει, από τα προβλήματά της. Μπορεί να μην έρθει καμία χώρα. Αυτό είναι ανοιχτό θέμα και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εκ των προτέρων, έτσι αφηρημένο, με αφηρημένο τρόπο. Θα σταματήσω εδώ, δεν ξέρω αν έπρεπε να προσθέσω κάτι άλλο. Μάρκο, ε, εκτιμώ ιδιαίτερα, λέει ο Μάρκο, την, ε, την ε, εντιμότητα, την ειλικρίνεια ε, είναι καλό που είχαμε αυτές ε, τις ε, συζητήσεις. Οι χώρες έχουν να κάνουν επιλογές όπως και οι οργανισμοί. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε κατάματα την πραγματικότητα. Θα ήθελα να κάνω μερικά γενικά σχόλια προτού περάσω σε ορισμένα θέματα. Συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα, εδώ έχουμε μια γενική αρχή αν θέλετε, πολύ γενική η άποψη ότι η δημοσιονομική πειθαρχία με δικαιοσύνη είναι αντινομία ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα και τα δύο να επιτευχθούν, αυτό είναι εσφαλμένο. Και το καλύτερο παράδειγμα στην Ευρώπη είναι οι χώρες του Βορρά, που είναι οι καλύτερες ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία και τα ταυτόχρονα εγγυώνται υψηλό επίπεδο δικαιοσύνης και ισόνομης διανομής των αγαθών. Έχουμε το θέμα του εισοδήματος και της ανάπτυξης. Έχουμε στην Ευρώπη μια δημοσιονομική στρατηγική που ε, δεν είναι μειώσεις παντού μη διαφοροποιημένο τρόπο. Το ΕΚΟΦΗΝ έχει θέσει ορισμένες αρχές για την δημοσιονομική πολιτική με τη σημερινή συγκυρία. Οι περισσότερες χώρες έχουν πολύ ψηλό χρέος και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την μείωση του χρέους. Οι δημοσιονομικές ε, πολιτικές θα πρέπει να είναι εξυγίανση, αλλά ταυτόχρονα ενώ ορισμένες ε, ευάλωτες χώρες δεν έχουν επιλογή, δεν, έχουν, ε, δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά αν δεν αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη. Άλλες χώρες έχουν περισσότερο περιθώριο ελιγμού και μπορούν να μειώνουν το έλλειμμα και οι σταθεροποιητές οι κανονικοί θα παίξουν το ρόλο τους. Υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική διαφοροποίηση ανάμεσα στις χώρες ε, και γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο αυτό την δημοσιονομική στάση στην Ευρώπη. Αποδίδουμε ιδιαίτερη ε, σημασία σε αυτό την ε, την μείωση των δαπανών, την συμπίεση, την δημοσιονομική. Όλες οι στρατηγικές δεν είναι οι ίδιες και στην ε, στρατηγική Ευρώπη 2020 οθούμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τις σωστές επιλογές ε, όσο προς την ποιότητα και τη σύνθεση. Είναι σαφές ότι οι χώρες, και εδώ υποστηρίζω πλήρως τον Κλάους, ότι οι χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα και άλλες ίσως, αυτές οι χώρες περνάνε πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Βεβαίως τα αποτελέσματα δεν πρέπει κανείς να δει αμέσως πλήρως, δεν μπορεί. Οι προϋποθέσεις για να αρχίσει και πάλι η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα πρέπει να διαμορφωθούν. Και αυτή είναι η περίπτωση της Ιρλανδίας κυρίως, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι είναι ένα πρόγραμμα που πέρασε όλο τον κύκλο και είναι περίπτωση της Λετωνίας ε, ήταν η πρώτη περίπτωση και εκεί όντως η χώρα πέρασε μια περίοδο προσαρμογής που ήταν πάρα πολύ σκληρή και μετά ανέκτησε την ανταγωνιστικότητα, μείωσε το έλλειμμα και το χρέος πέρασε σε πλεόνασμα και είχε ε, η ανάπτυξη πέρσι και τώρα οι προβλέψεις δεν είναι βεβαίως και ε, τόσο ε, αισιόδοξε, διότι υπάρχει ένας μαρασμό γενικό, αλλά η χώρα βλέπετε μπορεί να ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές και πολλές φορές πολύ πιο γρήγορα από ό,τι κανείς το περιμένει αρχικά. Ε, στη Λετωνία 100.000 μετανάστευσας Πού θα πρέπει να πάνε αυτές, αυτοί οι άνθρωποι. Στην Λετωνία 100.000 άτομα έφυγαν από τη χώρα σε μια χώρα που έχει κάπου κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια πληθυσμό. Αυτή είναι κινητικότητα και δεν είναι κακό αυτό. Τελειώσαμε. That in implementing, in implementing the program, we actually had to correct the initial intention of the of the government at the at the time and insist